Meine Damen Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους θερμά στην πρώτη συνεδρίαση μετά τις θερινές διακοπές. Βλέπω πολλούς συναδέρφους ε, που φαίνονται ξεκούραστοι ελπίζω τις διακοπές της, να τις ε, εκμεταλλευτήκατε ώστε να μαζέψετε δυνάμεις. Ε, κάποιοι βρίσκονται ακόμα σε διακοπές από ό,τι φαίνεται ή στο δρόμο ε, καθοδόν. νομίζω όμως ότι θα, πρέπει να ξεκινήσουμε για να εκμεταλλευτούμε και τον χρόνο μας για τις πολιτικές μας εργασίες. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχουν παρατηρήσεις για την ε, ημερήσια διάταξη. Κατ' εξαίρεση δεν έχουμε καμία τροποποίηση τη ημερήσια διάταξη. Α, ε, ο συνάδελφο Ρίβιχερ, ε, ήλπιζα ότι θα τη βγάλουμε χωρί τροποποίηση στην ημερήσια διάταξη. Ε, θα ξεκινήσει καλά το φθινόπωρο. Ήθελα να ρωτήσω μόνο την επόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη, ε, έχουμε συνεδρίαση μισή ημέρα. Ε, πότε έχουν προγραμματιστεί οι ψηφοφορίε. Διότι νομίζω ότι ε, συνήθω έχουμε τι ψηφοφορίε τη δεύτερη μέρα τη συνεδρίαση θα ήταν χρήσιμο καιρός, να γνωρίζουμε και τι θα βρίσκεται στη μέση διάταξη. Ε, πρόεδρος, ε, ναι, Έχουμε κάποιες πρώτες ενδείξεις, ε, δεν έχουμε όμως ε, όλες τις πληροφορίες ακόμα. Σας ευχαριστώ πάντως. Πάμε στις ανακοινώσεις του Προέδρου. Ε, μία... Ε, ε, μία έκκληση για ε, υποστήριξη. Έχουμε ε, φτιάξει το πρόγραμμα για τις συνεδριάσεις των συντονιστών της επόμενης χρονιάς. αλλά το Policy Department έχει εξετάσει αυτό και έχει αλλάξει κατά πολύ το πρόγραμμα και αυτό που πρόσεξα και που με ενοχλεί κάπως είναι ότι επανειλημμένα έχουν ε, αλλάξει τις συνεδριάσεις μας δεύτερα ε, Τρίτης σε Τετάρτη Πέμπτη και μάλιστα Πέμπτη απόγευμα. Ε, αυτό μπορεί να φαίνεται πολύ κανονικό, αλλά ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Και εγώ ξέρω τι σημαίνει αυτό και γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω να δώσουμε εντολή στη γραμματεία να ξανασυζητήσει με το Policy Department ώστε τουλάχιστον να αλλάξουν κάποιες από τις ημερομηνίε αυτές διότι ε, τις προτάσεις μας εμείς τις κάναμε μετά από καλό συλλογισμό και ε, πιστεύουμε ότι ε, η λύση που μας προτείνουν δεν είναι πολύ ε, σωστή. Το να αλλάξουμε καμιά δυο φορές από Δευτέρα, Τρίτη σε Τετάρτη, Πέμπτη μπορεί να μην πειράζει, αλλά το να γίνεται αυτό συνέχεια και μάλιστα να έχουμε συνεδρίαση Πέμπτη απόγευμα, αυτό δεν είναι πολύ καλό, πόσο μάλλον που συνήθως Πέμπτη απόγευμα οι συνεδριάσεις είναι μάλλον light, είναι κάπως συνεδριάσεις όχι πολύ σημαντικές. Ε, δεν βλέπω να υπάρχει καμιά αντίρρηση. Ε, παρακαλώ λοιπόν να με υποστηρίξετε ώστε να μπορέσουμε να ε, αλλάξουμε πάλι το πρόγραμμα ώστε να μην ε, χρειασ... χρειαστεί ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις εργασίες μας. Προχωράω λοιπόν στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Φοντέιν, πρόεδρο της Μπέρεκ, ο οποίος θα μας κάνει μια παρουσίαση. Ε, των δραστηριοτήτων ε, του Μπέρεκ. Κατόπιν θα δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν. που θα μας ε, παρουσιάσει το θέμα της περιαγωγής και θα ζητήσουμε από τον κύριο Φοντέιν να μας παρουσιάσει τις θέσεις του για το θέμα αυτό και κατόπιν θα έχουμε συζήτηση, εφόσον συμφωνείτε. Έχουμε χρόνο. Θα ήταν όμως χρήσιμο ε, να συζητήσουμε μαζί τα δύο θέματα αυτά. Ξεκινάμε λοιπόν με την ε, παρουσίαση του κυρίου Φοντέιν, ε, Προέδρου του Μπέρεκ, που θα μας παρουσιάσει τις δραστηριότητες του Μπέρεκ. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω τον κύριο Φοντέιν και όχι κύριο Μπέρεκ, όπως είπα κατά λάθος, συγγνώμη. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και σας δίνω το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ήτρε, <laughs> απαντά κύριε Σποντέιν. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Εκ μέρους της Μπερέκ και προσωπικά σας ευχαριστώ και για την πρόσκλησή σας ως προεδρεύοντες, συνδυασμένοι προεδρεύοντες των ρυθμιστικών αρχών, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να έχουμε μια τακτική επαφή με το Κοινοβούλιο, με την Επιτροπή και το Συμβούλιο και ελπίζω και στο μέλλον να συνεχιστεί αυτό. Πρώτα θα ήθελα να σας παρουσιάσω μια περίληψη της ετήσιας έκθεσης για το 2010 και των εργασιών τις οποίες αναλάβαμε για το 2011. Είμαστε μια νέα οργάνωση, παρόλα αυτά προχωράμε. Ε, σήμερα μετά από την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα σας παρουσιάσω και τις βασικές συστάσεις ε, της ε, Μπερέκ για την αναθεώρηση του κανονισμού roaming. Αυτό είναι πάρα πολύ θα έλεγα σωστά χρονισμένο γιατί χθε εμείς δημοσιεύσαμε ε, την, ε, τις συστάσεις μας για την αναθεώρηση της πρότασης για την περιαγωγή. Το 2010 στην ετήσια έκθεση η οποία είναι εκρήθη τον Μάιο του 2011 η Μπερέκ ε, λειτουργήσε υπό την προεδρία του Τζον Ντόχερτη του Ιρλανδού συναδέλφου. Ξέρετε ότι ήταν ένα έτος το πρώτο έτος μάλλον της λειτουργίας δέθηκαν τα θεμέλια της Μπερέκ η οποία λειτουργεί πλήρως φέτος. Πολλές λοιπόν από τις προηγούμενες μας δραστηριότητες ήταν ματαβατικές σε σχέση με τη συγκεκριμένη οδηγία πλαίσιο και ακολουθήσαμε επίσης και αυτά τα οποία είχε κάνει η ομάδα των ρυθμιστικών αρχών η προκάτοχος της Μπερέκ. Τρεις δρόμους στην ουσία ακολουθήσαμε. Η οργάνωση, είναι ο ένας, οι προκλήσεις το δύο και οι αλλαγές στο πλαίσιο το τρία, ο τρίτος δρόμος. Αυτά συνεχίζουμε και, συνεχίσαμε και θα συνεχίσουμε μάλλον και στο τέλος του έτους, μέχρι το τέλος του έτους. Δύο σημαντικά θέματα στην εναρμόνιση τα οποία αντιμετωπίσαμε το 10 ήταν η διεθνής περιαγωγή. Θα αναφερθώ στην σειρά των ενεργειών μας πέρυσι και φέτος και Επίσης ε, και το NGA, ε, οι προσπάθειες για την πρόσβαση νέας γενεάς ε, που έχουμε αρχίσει εδώ και αρκετό καιρό. Αναφερθήκαμε στην υπαγωγή της λειτουργίας των ρυθμιστικών αρχών στην υπάρχουσα διάταξη και στην πιθανότητα διεύρυνση αυτής της ρύθμισης. Αυτή η σύσταση είναι η βάση της ανάλυσης που θα παρουσιάσω αργότερα και προτείνει βλέπει μάλλον διαρθρωτικά προβλήματα στην αγορά. Αναφέρουμε ότι με αυτές τις διαρθρωτικές αλλαγές οι τιμές θα συνεχίσουν να σταματούν σε συγκεκριμένα επίπεδα χωρίς πιθανότητες περαιτέρω μειώσεων. Τα βασικά θέματα που επίσης συζητήσαμε είναι σχετικά με τις αποφάσεις που ελήφθησαν το 10. Δημοσιεύσαμε μία έκθεση με ένα instantane θα έλεγα της εικόνας που παρουσιάζει η χρήση του roaming της περιαγωγής προς τους καταναλωτές και μια επίσημη επίσης σύσταση σχετικά με τις συστάσεις για τις προσβάσεις νέας γενεάς, συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι τροποποιημένες αυτές συστάσεις έγιναν δεκτές το μήνα Δεκέμβριο. Δεύτερον, οι αναδυόμενες προκλήσεις, καταρχάς η σύγκληση όπως γνωρίζετε και η ουδετερότητα του δικτύου είναι κάτι το οποίο παραμένει πάντα προτεραιότητα. Για τις συγκλήσεις η Μπερέκ δημοσίευσε μια έκθεση για την παροχή ε, ευρέως δικτύων και κάναμε και μια ανάλυση των ε, αυτό του τύπου των δικτύων και ε, είδαμε πώς εξελίσσονται όλα αυτά στις τηλεπικοινωνίες πρόσφατα τον Ιούνιο του 10. Η Μπερέκ δημοσίευσε επίσης ε, μια παρουσίαση της σημερινής κατάστασης στα πλαίσια της καθολικής υπηρεσίας υπογραμμίζοντας τις διάφορες εθνικές στρατηγικές που έχουν σαν στόχο την εξέλιξη και ε, διάταξη θα έλεγα της, του ευρέως φάσματος που απαιτεί περαιτέρω προσοχή είναι ένα θέμα το οποίο παραμένει πάρα πολύ σημαντικό στα πλαίσια των προτεραιοτήτων της ΜΠΕΡΕΚ. Η συζήτηση για την ευετερότητα των δικτύων, όπως γνωρίζετε, έχει εντατικοποιηθεί το 2010. Απαντώντας στις διαβουλεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρατηρήσαμε σαν Μπερέκ ότι εμείς δεν έχουμε δει μέχρι τώρα πολλά προβλήματα και τα περισσότερα από τα προβλήματα αυτά ελήφθησαν χωρίς περαιτέρω θεσμικές παρεμβάσεις. Πράγματι οι διατάξεις του αναθεωρημένου δικτύου πλαισίου είναι στόχος και των εργασιών μας το 2011. Ξέρετε ότι έχουν υπάρξει πολλές εξελίξεις στον τομέα αυτό και στην Ολλανδία, στη χώρα μου. Το τρίτο πλαίσιο εργασίας μας είναι το ρυθμιστικό θεσμικό πλαίσιο. Βασικό στόχος της Μπερέκ ήταν να δημιουργήσει το λεγόμενο Berek Office στη Ρήγα. Αποφασίστηκε το 2010. Το προσωπικό ε, αυξάνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα και ελπίζουμε να έχουμε 20 ε, μέλη που θα εργάζονται στο γραφείο μας στη Ρήγα μέχρι το τέλος του χρόνου. Οκτώ εργάζονται ήδη και είναι ε, έτοιμοι να δεχθούν την πρώτη επίκληση αναφοράς του άρθρου 7. Ε, βρήκαμε χώρο γραφείων, περιμένουμε να αυτονομηθεί το γραφείο και να ε, εκινήσει επίσημα τον Οκτώβριο. Ε, ελπίζω να σας συναντήσω όλους στη Ρήγα όταν έχουμε τα εγγένεια. Με την δημιουργία του γραφείου Μπέρεκ δημιουργήσαμε κάποιες νέες διαδικασίες. Η πιο σημαντική είναι η διαδικασία άρθρου 7 και 7α Επί τη βάση λοιπόν των άρθρων 7 και 7α εμείς θα πρέπει να αναθεωρούμε τις αποφάσεις S&P που λαμβάνονται από, τους μεμονωμένους, από τις μεμονωμένες ρυθμιστικές αρχές. Και στην ουσία πρόκειται και για μία θα έλεγα αξιολόγηση ομολόγων, ομολόγων υπηρεσιών ρυθμιστικών αρχών και προσπαθούμε να δούμε αν όλα γίνονται σε σωστό επαγγελματικό επίπεδο. Περιμένουμε τις πρώτες επικλήσεις σύντομα, υπήρξε μία πρώτη πριν από την εισαγωγή του πλαισίου, αλλά περιμένουμε τις πρώτες επίσημες ε, σύντομα και θα παρακαλουθήσουμε προσεκτικά τα άρθρα της διαδικασίας του άρθρου 7 και θα αναφερθούμε σε αυτά τακτικά. Θα περάσω τώρα στο 2011. Το πρόγραμμα εργασίας μας για το 2011 οργανώθηκε επί τη βάση των τριών ιδίων δρόμων θα έλεγα που ακολουθήσαμε το 10 δηλαδή εναρμόνιση, αναδιόμενες αγορές και νέο πλαίσιο μπερέκ. Θα αναφερθώ μόνο σε ορισμένα θέματα τα οποία θεωρώ πιο κρίσιμα. Καταρχάς η προσπάθεια που κάνουμε για την περιαγωγή θα επανέλθουμε σε αυτή. Παρακολουθούμε συστηματικά τις εξελίξεις στην αγορά περιαγωγής και σε επίπεδο χονδρικής αγοράς και σε επίπεδο λιανικής. Επί τη βάση αυτού του ελέγχου και της αναλύσεως που δημοσιεύσαμε πέρυσι, εκδώσαμε και τις συστάσεις μας για την αναθεώρηση του κανονισμού περιαγωγής. Θα επανέλθω σε αυτά αργότερα. Δεύτερον, η ουδετερότητα του δικτύου για μας είναι βασική μας προτεραιότητα. Θα εξακολουθήσουμε να ασχολούμεθα με θέματα συγκεκριμένα όπως η διαφάνεια, η ποιότητα και οι διακρίσεις. Πιστεύουμε ότι θα ξεκινήσουμε μια δημόσια διαβούλευση τον μήνα Οκτώβριο για θέματα διαφάνειας σχετικής με την ουδετερότητα των δικτύων. Η προσπάθεια που κάνουμε για την ποιότητα παροχής υπηρεσίας και για τις διακρίσεις θα είναι έτοιμη για δημοσίευση τον μήνα Δεκέμβριο. Ένα, μια άλλη βασική προτεραιότητα είναι η προσπάθεια την οποία κάνουμε σχετικά με το ευρύ δίκτυο και τα δίκτυα επόμενης γενεάς. Συνεργαζόμαστε στα πλαίσια μια ανάλυση σε βάθος των μέσων που χρησιμοποιούν οι κυβερνήσει και οι εμπλεκόμενε αγορέ για την βελτίωση τη σωστή χρήση του ευρέως φάσματο. και θα χρησιμοποιήσουμε τις παρατηρήσει μα αυτέ, τις συστάσει που θα κάνουμε για τη χρήση αυτού του μηχανισμού. Ταυτόχρονα εμείς αναφερόμεθα και στην λογιστική των ρυθμιστικών μέτρων σχετικά με τα δίκτυα επόμενης γενιάς. Και για τα θέματα αυτά, όπως είπα, θα ξεκινήσουμε με δημόσιες διαβουλεύσεις. Υπάρχει μια μικρή αλλαγή σχετικά με το τι κάναμε ανάμεσα στο 10 και αυτό που κάνουμε στο 11. Δίδουμε ακόμα περισσότερη προσοχή στην, στην συνοχή θα έλεγα των μέσων τα οποία χρησιμοποιούμε για να διορθώσουμε τα προβλήματα. Αναλύσαμε την εφαρμογή των κοινών θέσεων των ρυθμιστικών αρχών σχετικά με τα δίκτυα χονδρικής τα οποία ακόμα δεν έχουν απελευθερωθεί. Πιστεύουμε ότι η αναθεώρηση των κοινών θέσεων θα πρέπει να γίνει γρήγορα και η αναθεώρηση αυτή θα πρέπει νομίζω να οδηγήσει, αυτό είναι ο στόχος μας, σε περαιτέρω εναρμόνιση, σε αυξημένη εναρμόνιση. Όπως είπε η κυρία Νέλη Κρός, αυτό δεν είναι ε, για να δημιουργήσουμε ένα μέγεθος κοινό για όλους, ένας κανόνας που να ισχύει για όλους. Αλλά από την άλλη δεν λέμε ότι χρειάζονται και 27 μεγέθη για κάθε μία χώρα της Ευρώπης. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να βρούμε τη μέση οδό ένα άλλο τομέα τη δραστηριότητας της ΜΠΕΡΕΚ, τον οποίο βρίσκω πολύ σημαντικό, είναι οι σχέσεις μας με τις μπλεκομένους στην αγορά. Είδατε ότι αναφέρθηκα πολλές φορές σε δημόσιες διαβουλεύσεις, το κάνουμε όσο μπορούμε, είναι τακτικό τμήμα της προσπάθειάς μας και μας δίδουν πράγματι εξαιρετικέ πληροφορίες από πλευράς των εμπλεκομένων συμμετεχόντων στην αγορά, των καταναλωτικών οργανώσεων κτλ. Ως προεδρεύων τους Μπερέκ προσπαθώ εγώ να είμαι σε επαφή συνεχώς με τους εμπλεκομένους και κερδίζω πάρα πολύ από αυτό, συμμετέχω σε σεμινάρια, συνέδρια κτλ. Ε, δέχομαι προκλήσεις από την Έτνο και την Έκτα, από, το, από τον Διεθνή Δικηγορικό Σύλλογο και από μεμονωμένες ρυθμιστικές αρχές. Εν πάση περιπτώσει οδηγούμε τώρα στο κλείσιμο της σύντομη παρουσίασής μου πράγματι στα πλαίσια της Μπερέκα να εξελίσσουμε το στρατηγικό μας πρόγραμμα για τα επόμενα χρόνια. Προσπαθούμε να δούμε στο μέλλον πέραν του ενός ή δύο ετών. Ήδη κάναμε για το θέμα αυτό μια συνεδρίαση του Δικητικού Συμβουλίου. Θα χρησιμοποιήσουμε πλήρως τα γραφεία της Ρήγα τον επόμενο μήνα. Θα δούμε ποια θα είναι η στρατηγική την οποία θα ακολουθήσουμε. Συμπερασματικά λοιπόν θα έλεγα ότι η Μπερέκ έχει ε, ε, έμπειρα μέλη στο εσωτερικό της αλλά είναι μια νεαρή εισαγωγικά οργάνωση η οποία πρέπει να αποδείξει ότι είναι χρήσιμη. Το 2010 ε, η Μπέρεκ στην ουσία συνέχιζε αυτά που έκανε η προκάτοχος οργάνωση, η ERG. Μαντουρέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Φοντέιν και για την παρουσία του εδώ, αλλά και για το έργο του φορέα σε ό,τι αφορά την πρόταση περιαγωγής. Και τον ευχαριστώ για την έκθεσή του που θα μας ε, βοηθήσει σίγουρα πολύ στο έργο μας. Και μια και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ τον κύριο Φοντέν, θα ήθελα να να αξιοποιήσω την ευκαιρία και να υποβάλω κάποιες ερωτήσεις. Από τη δημιουργία του φορέα πέρασε λίγο χρονικό διάστημα. Θα ήθελα να θέσω συγκεκριμένες ερωτήσεις για τη λειτουργία του φορέα αυτού. Μας μιλήσατε για τις λειτουργίες του φορέα, του Μπερέκ. Και από ό,τι θυμάμαι από τις συζητήσεις που είχαμε, που κατέληξαν στην ίδρυση του Μπερέκ, θυμάμαι ότι το ζητούμενο ήταν να γίνει ο φορέας αυτός, ο Ευρωπαϊκός Φορέας, ένα σώμα που θα εξασφαλίζει ένα σημαντικό βαθμό ανεξαρτησίας. Αυτό, αυτή ήταν η επιθυμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ερωτώ λοιπόν, πιστεύετε ότι ο Μπερέκ ανταποκρίνεται πλήρως αυτές τις επιθυμίες του Κοινοβουλίου ως προς την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας του ποια η σχέση του Μπερέκ ε, και απέναντι στην Επιτροπή αλλά και απέναντι στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Δεύτερη ερώτηση. Εσωτερική λειτουργία του Μπερέκ και ιδιαίτερα λειτουργία του σε σχέση με τον κανονισμό. Είπατε ότι εν γέννη είστε ικανοποιημένοι από το ρυθμιστικό πλαίσιο του κανονισμού. Ερωτώ αν έχετε σχόλια ή παρατηρήσεις ή προτάσεις βελτίωσης του κανονισμού εν των επικείμενων αναθεωρήσεων. Και τρίτη και τελευταία ερώτηση. Πιστεύετε ότι ο Μπερέκ είναι αποτελεσματικό εργαλείο προκειμένου να μειωθούν τα χάσματα στις προσεγγίσεις των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Γιατί είπατε ότι απότερο στόχος είναι η υλοποίηση της ενιαίας αγοράς. Πιστεύετε ότι μεσοπρόθεσμα θα έχουμε μια γνήσια ενιαία αγορά για τις ηλεκτρονικές ε, επικοινωνίες. Η κυρία Τόγια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να χαιρετήσω και εγώ τον Προεδρεύοντα της Μπερέκ. Το ε, ερώτημά μου έχει σχέση με την τελευταία παρατήρηση της Τερέσα Μαντουρέλ σχετικά με το ρόλο που μπορεί να έχει η Μπερέκ για να μειωθούν οι διαφορετικές εθνικές πραγματικότητες, να έρθουν πιο κοντά, γιατί εμποδίζουν την δημιουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Λαμβάνω υπόψη ότι η δραστηριότητα στην οποία αναφερθήκατε αναφέρεται σε μια πολύ σύντονη χρονική περίοδο, αλλά διαρωτώ με αν η διαδικασία την οποία προβλέψατε σχετικά με την αναφορά στο 7 και στο 7α είναι αποτελεσματική και στα πλαίσια της αξιολόγησης ομολόγων είναι μια ευγενική αμοιβαία εξέταση θα έλεγα ανάμεσα σε ισότιμους εταίρους η οποία δεν επιτρέπει στην ΠΕΡΕΚ να παρεμβαίνει εκεί όπου διαπιστώνει όπου οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δεν λειτουργούν σωστά ή δεν είναι ανεξάρτητες για πολιτικούς λόγους ή εν πάση περιπτώσει δεν είναι επαρκής αρκετά οι αρχές αυτές και δεν μπορούν να φέρουν εις πέρα σε αυτό το οποίο καλούνται να κάνουν. Διαφορετικά στοιχεία υπάρχουν σε κάθε χώρα, υπάρχουν πολλές φορές ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και τον επιχειρηματικό κόσμο πολλές συμπτώσεις και αντιθέσεις συμφερόντων και γι' αυτό το σημείο ισορροπίας το οποίο έχετε καταλήξει στο σημείο 7 με το άρθρο 7 πιστεύετε ότι είναι ικανοποιητική. Εγώ θα προτιμούσα να έχω μια Ευρωπαϊκή Αρχή πολύ ισχυρότερη από τις εθνικές αρχές αντίστοιχες. Βέβαια επαναλαμβάνω η περίοδος στην οποία δραστηριοποιηθήκατε είναι πολύ πολύ σύντομη. Ευχαριστώ Παύλο Ρίμπιχ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να, συγχαρώ, να σας συγχαρώ για το νέο ξεκίνημα. Πιστεύω ότι είναι αποφασιστική σημασία η ε, ερώτησή μου έχει να κάνει με τα δίκτυα της επόμενης γενιάς. Τι γίνεται εκεί με την ουδετερότητα του δικτύου. Θα υπάρχει ε, διαφορά ανάμεσα στα ε, παρόντα συστήματα κινητών τηλεφώνων και του δικτύου νέας γενιάς και πώς θα τεθούν τα πρότυπα και πιστεύετε ότι είναι δυνατόν να έχουμε διασυνοριακές διατάξεις ώστε να μπορούν τα δίχτυα αυτά να χρησιμοποιηθούν από όλου όσου ενδιαφέρονται. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφο Λάμπερτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα μιλήσω αγγλικά κύριε Φοντέιν. Καταρχήν θα ήθελα να ε, συμφωνήσω με την ερώτηση του Ολλανδού συναδέρφου σχετικά με την ουδετερότητα των δικτύων, διότι από τη μία είπατε ότι υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις που μπορούσαν να λυθούν χωρίς ε, ρυθμιστική παρέμβαση χωρίς νομοθετική παρέμβαση και μάλιστα κάποια κράτη-μέλη σχεδιάζουν να αναλάβουν μέτρα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, διότι εσείς είπατε ότι εσείς ε, χρησιμοποίησατε την ε, λέξη εναρμόνιση, την οποία χρησιμοποιούν λίγοι ε, σήμερα. Η κυρία Τόγια είπε ότι ο φορέας Μπέρεκ δεν έχει την εξουσία να εφαρμόσει, να επιβάλλει ρυθμίσεις. Ωστόσο, εσείς μιλήσατε για εναρμόνιση. Και η δεύτερη μου ερώτηση συνδέεται με αυτό. Πιστεύω ότι είναι έγκυρα αυτά που λέτε, αλλά πόσο συμφωνούν με αυτά ε, τα άλλα μέλη του Συμβουλίου. Ε, τα κράτη-μέλη πιστεύουν ότι πρέπει να επιδιώξουμε μια ε, ε, εναρμόνιση από τη βάση προς τα πάνω ε, σε όλους τους τομείς που αναφέρατε συμπεριλαμβανομένοι στη ουδετερότητας του δικτύου ή πιστεύετε ότι είσαστε πιο προοδευτικός στο θέμα αυτό σε αντίθεση με κάποιους άλλους που μπορεί να επιθυμούν μάλλον μια καθυστέρηση. ήθελα να ακούσω τη δική σας θέση, πώς πιστεύετε ε, ότι έχουν τα πράγματα, διότι ως πράσινοι και, ε, και πολλοί άλλοι εδώ μέσα ε, θέλουν εναρμόνιση των δικτύων και εξάλληψη των συνόρων στο θέμα αυτό. αυτά που, που λέτε είναι πολύ ευχάριστα για μας. Ήθελα όμως να ξέρω κατά πόσο συμφωνούν με αυτά και οι συνάδελφοί σας. Ευχαριστώ η συνάδελφος Χέρτσοκ. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τον ε, πρόεδρο του Μπέρεκ. Μία γενική παρατήρηση ή ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Η ευρωπαϊκή αγορά πόσο ενωμένη είναι. Κάποιες αγορές έχουν μείνει πίσω, κάποιες ε, έχουν πολλές ιδιαιτερότητες. Η Ευρώπη είναι εξίσου διχασμένη στο θέμα αυτό όσο και σε άλλα ερωτήματα. Μπορείτε να απαντήσετε στο θέμα αυτό. Τελευταία που ζητάει το λόγο είναι η συνάδελφος Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για τις πληροφορίες που λάβαμε. Ε, ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπαν ήδη άλλοι συνάδελφοι που έχουν να κάνουν με την ε, ουδετερότητα των δικτύων. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ουδετερότητα των δικτύων, ε, ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να υπάρχει κάλυψη κατά 100% για τις ευρυζωνικές συνδέσεις. Θα ήθελα να αναφερθώ σύντομα ε, στην νομοθετική ρύθμιση για την περιαγωγή, αν και από ό,τι κατάλαβα θα το συζητήσουμε αυτό στη συνέχεια. Η ε, νομοθεσία αυτή ε, εισήχθη επειδή δεν λειτουργούσε πολύ καλά η αγορά. Γι' αυτό το 2009 είδαμε τη σχετική νομοθεσία. Η Κομισιόν κατόπιν υπέβαλε πρόταση στο μέλλον οι τιμές για τα μηνύματα σε κινητό, τα SMS και για ε, την διαβίβαση δεδομένων ε, για τις τιμές αυτές να υπάρχει κάποια οροφή. Και οι τιμές να διαμορφώνονται ανάλογα με αυτές ε, των ε, εθνικών δικτύων. Μιλάμε για εσωτερική αγορά και γι' αυτό οι τιμές περιαγωγή δεν θα πρέπει να είναι πιο ψηλέ από τις ε, εθνικές τιμές. Ε, θα ήθελα πολύ να ακούσω την ε, άποψή σας. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στον κύριο Φοντέιν για να απαντήσει. Thank you. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Δελκαστήγιο καταρχήν για τα ευγενικά της λόγια. Δεν ξέρω αν από αυρότητα θα έπρεπε να απαντήσω Ολλανδικά στον κύριο Νίστερ. Φοβάμαι, δεν ξέρω τι ήθιστε εδώ, αλλά φοβάμαι ότι αν του μιλήσω Ολλανδικά κανένα δεν θα καταλάβει. Προτιμώ να απαντήσω στα Αγγλικά. Ε, Αυτά τα θέματα που αναφέρετε είναι πολιτικά και εμεί στον Μπερέκ δεν είμαστε πολιτικοί. Είναι κάπω πρόημο να σχολιάσουμε μόνο με ένα θέματα εθνικών οθεσιών ενώ συνεχίζονται οι έρευνες. Από δικές μας έρευνες και μελέτες διαπιστώσαμε ότι σε ό,τι αφορά τα θέματα διαφάνειας και την ιδιαιτερότητα ο κόσμος ξέρει, ε, θα πρέπει να ξέρει τι αγοράζει και γιατί πληρώνει. Αυτή είναι η βασική αρχή. Και αυτή θα πρέπει να είναι η κρατούσα αρχή. Πάντως, ε, μερικές δράσεις ε, ίσως είναι πρώιμες από κάποιες εθνικές νομοθεσίες, αλλά δεν θα ήθελα να σχολιάσω εγώ τέτοιες νομοθετικές ε, εθνικές πρωτοβουλίες. Στην Ευρώπη, εμείς με το φορέα μας, το Μπερέκ, ε, προσπαθούμε να μην εμπλακούμε σε πολιτικά ζητήματα, απλώ να μελετήσουμε και να ερευνήσουμε τα επίκαιρα προβλήματα, τα τεχνικά ζητήματα που ανακύπτουν. Και αν θέλουμε το διαδίκτυο να είναι ανοιχτό ένα ανθρώπινο δικαίωμα για όλους ή αν θα πρέπει να υπάρχει κάποιος περιορισμός, αυτό είναι μια πολιτική επιλογή. Πάντως θα πρέπει τουλάχιστον στην Ευρώπη να έχουμε μια μειόμορφη προσέγγιση. Αλλά αυτό είναι θέμα πολιτικών και όχι ρυθμιστών. Εμείς θα δώσουμε συμβουλές στους ε, νομοθέτες για τις συνέπειες που θα έχουν δεδομένες αποφάσεις στην αγορά. Και δεν θα ε, ακολουθούμε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η μόνη κατεύθυνση που ακολουθούμε είναι ότι στην Ευρώπη η συζήτηση δεν ήταν τόσο οξύ όπως στις Ηνωμένε Πολιτείε και δεν είχαμε τόσο οξέα προβλήματα όπως σε άλλες χώρες του κόσμου και άλλες περιοχές του κόσμου. Κύριε Μαντουρέλ, μίλησατε για την ανεξαρτησία του Μπέρεκ. Νομίζω ότι το θέμα της ανεξαρτησίας ε, είναι πραγματικά ε, σημαντικό, νευραλγικό. Βέβαια ξέρετε ότι έχουμε 27 ε, μέλη παρατηρητές στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μπερέκ, προσώπους των ε, χωρών μελών και στο Κοινοβούλιο έγινε μακροχρόνια συζήτηση για το κατά πόσο οι εξουσίες του άρθρου 7 θα πρέπει να δίνονται περισσότερο στους ρυθμιστές, στις ρυθμιστικές αρχές ή στην Ευρώπη με ένα πιο κεντρικό τρόπο. Και γνωρίζουμε ότι υπάρχει αρκετή επιφυλακτικότητα και σκεπτικισμό. Πάντως στις συνεδριάσεις μας εμείς έχουμε επίγνωση αυτού του γεγονότος και γνωρίζουμε ότι αν εμεί ως Μπερέκ δεν δείξουμε ότι είμαστε επαγγελματικοί, ανεξάρτητοι και ικανοί απέναντι ε, στου πολιτικού στην Κομισιόν, απέναντι ε, σε όλου. αν δεν αποδείξουμε αυτή την ανεξαρτησία και τον επαγγελματισμό προ την εντολή μα, θα υποστούμε δερμήτατε κριτικέ. Και στην πρώτη αναθεώρηση θα γίνουν αλλαγέ. Αυτό θα ήθελα να σας πω ότι και εγώ και οι συναδελφοί μου έχουμε πλήρη συνείδηση του ότι τα μάτια είναι στραμμένα πάνω μας ε, και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις διαδικασίες του άρθρου 7, στην ανεξαρτησία και παρακολουθούμε κριτικό ε, μάτι τις ε, συμβουλές που θα δώσουμε, τις γνωμοδοτήσεις γιατί διαπίστωσα ότι πολλές ερωτήσεις περιστράφηκαν γύρω από το ίδιο θέμα αν θα αρκέσει αυτή η αναθεώρηση ισοτήμων στα πλαίσια της διαδικασίας 7. Πάντως είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι όσοι ζήτησαν αλλαγές στον κανονισμό, πιστεύω ότι στην πρώτη σκηνοποίηση του άρθρου 7 η λιδία λήθος για μας θα είναι αν ε, η πλειοψηφία των δύο τρίτων που έχουμε τώρα, που είναι όμω μια εσωτερική διαδικασία, αν θα χρειαστούμε αυτή την πλειοψηφία των δύο τρίτων και για την γνωμοδότηση. Γιατί είναι πολύ ενισχυμένη αυτή η πλειοψηφία. Θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε ικανοί να συγκεντρώσουμε την πλειοψηφία των δύο τρίτων για κάτι που ίσω είναι επικριτικό για ορισμένου συναδέλφου που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και αυτή θα είναι για μα η λιδία λήθο. Γιατί πολλέ κοινοποιήσει που έγιναν πριν το πλαίσιο Άνοικα ε, σε προηγούμενη κατάσταση. Τώρα θα περιμένουμε την πρώτη κοινοποίηση με το πλαίσιο και αν υπάρξουν εκεί προβλήματα και σίγουρα θα υπάρξουν και επίμαχες κοινοποίησεις και προς την Επιτροπή, θα υπάρξουν αμφιβολίες, θα πρέπει να γίνουν σοβαρές έρευνες, θα πρέπει να αποδείξουμε τον επαγγελματισμό μας και ότι μπορούμε να είμαστε επικριτικοί απέναντι στους ισοτήμους μας και ότι μπορούμε να συγκεντρώσουμε την πλειοψηφία των δύο τρίτων με επαγγελματισμό. Η μόνη διαβεβαίωση που μπορώ να σας δώσω είναι ότι οι συνάδελφοι στον ΠΕΡΕΚ έχουν απόλυτη επίγνωση ότι αν δεν ανταποκριθούν στο έργο τους θα υποστούν δρυμύτα τις κριτικές. Αυτό το γνωρίζουμε, έχουμε απόλυτη συνείδηση. Και θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τις, τροπολογι... τις κοινοποίησεις του άρθρου 7 και αν ε, η πλειοψηφία των δύο τρίτων θα δημιουργήσει πρόσκομα ιδιαίτερα όταν ε, υποβάλλεται μια γνωμοδότηση επικριτική. Πάντως είναι κάπως πρόημο να τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Ε, θέσατε ρωτήσει και για την ε, ενιαία αγορά, για την εσωτερική αγορά. Όπως είπα και στην εισαγωγή μου, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ενιαία λύση για όλους, γιατί υπάρχουν πραγματικά πολλές διαφορές δημογραφικές, γεωγραφικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει, πιστεύω, τις ίδιες μεθόδους που εφαρμόζονται από μια ρυθμιστική αρχή σε συγκεκριμένες ε, συνθήκες, να τις συγκρίνουμε με παρόμοιες συνθήκες. Αλλά πολλές φορές υπάρχουν διαφορές και στις υποδομές και οι λύσεις μπορεί να είναι διαφορετικές. Σε περίπτωση που έχουμε ίδιες περιστάσεις θα πρέπει να συγκρίνουμε παρόμοια εφαρμογή των ίδιων μέτρων. τέθηκε και μία ερώτηση για την αποτελεσματικότητα του σημείου 7 και ίσως ε, ε, μια κολακία προς τους ε, πολιτικούς. Θα πρέπει να δείξουμε, να αποδείξουμε μάλλον, δεν έγινε ακόμη αυτό, αλλά πολλές συζητήσεις έγιναν για το τι περιμένουν από εμά. Εμείς γνωρίζουμε ότι αν απλώς λέμε στους πολιτικούς αυτά που θέλουν να ακούσουν, δεν πρόκειται να μακροημερεύσουμε στο ΜΕΡΕΚ. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πίεση από τους ομότιμους, ε, γνωρίζουμε ότι μία από τις αδυναμίες αλλά και μία πρόκληση για μας είναι ακριβώς αυτή η πίεση και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γνωρίζουν ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτή η πίεση των νομοτήμων γιατί θέλουμε να καταλήξουμε σε κοινέ θέσει και αποκρισταλωμένε σαφεί αποφάσει στα πλαίσια του έργου μα στο άρθρο 7. Κύριε Ρουμπίχ, δεν μπορώ να σα δώσω μονοσήμαντη απάντηση. Ο Μπερέκ δεν ασχολείται με θέματα προδιαγραφών και προτυποποίησης. Εμείς είμαστε ρυθμιστική αρχή της αγοράς μιλήσαμε για την ενίσα και τα θέματα ασφάλειας και τα τεχνικά. Ίσως στο μέλλον ενισχυθεί και αυτή η πτυχή μας, αλλά αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε σε αξιολογήσεις της αγοράς και των ρυθμιστικών μέτρων προκειμένου να λειτουργεί εύρυθμα η αγορά. Φοβάμαι λοιπόν ότι δεν μπορώ να σας δώσω σαφή απάντηση. Κύριε Λάμπερτ, εγώ πολύ συχνά χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη που ξεκινά από H. Αυτό δεν είναι. Αυτή η λέξη, ε, harmonization, εναρμόνιση, πιστεύω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ευφύ τρόπο ε, υπό ε, τις σωστές περιστάσεις. Ο Μπερέκ είναι επαγγελματικός φορέας και όχι πολιτικός φορέας και από αυτή την άποψη έχει ένα σαφή ρόλο να καθορίσει μια πορεία. Γιατί πολύ συχνά η πορεία έχει οικονομικό περισσότερο χαρακτήρα παρά πολιτικό. Ευελπιστώ ότι ο Μπερέκ, οι συνάδελφοι αλλά και ο διαδοχός μου θα βρουν το σωστό ρόλο και θα δίνουν ε, τις συμβουλές ακόμη και όταν δεν ερωτώνται και προς το Συμβούλιο και προς την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο για την κατεύθυνση που κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Φυσικά υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή μεταξύ ε, του πολιτικού έργου και του τεχνικού επαγγελματικού Μερικέ φορές. Πιστεύω πάντως ότι ακόμη και αν παραβούμε μερικές φορές αυτή τη λεπτή γραμμή, ε, δεν πειράζει. Κύριε Χέρτσοκ, ρωτήσατε αν είναι ενοποιημένη η εσωτερική αγορά. Στις τηλεπικοινωνίες η απάντηση είναι ότι πόρα απέχουμε ακόμη. Πολιτικά και τεχνικά ναι, αλλά στην ουσία έχουμε τόσα πολλά εμπόδια στην εσωτερική αγορά που ο Μπέρεκ ε, χρειάζεται να αντιμετωπίσει σοβαρές προκλήσεις για να τα εξαλείψει. Ένα από αυτά είναι και το θέμα της περιαγωγής. Ε, κυρία Τσικάου, είπατε ότι η ουδετερότητα είναι σημαντική. Εμείς θέλουμε να επικεντρωθούμε στην οικονομική πρακτική συζήτηση, να ξεφύγουμε κάπως από μια πολλωμένη, πολλές φορές πολιτική συζήτηση. Στο θέμα της παραγωγής θα επανέλθουμε αργότερα. Είναι το δεύτερο θέμα που θα εξετάσουμε σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περιαγωγή. Τώρα, την επιθυμία μείωση του κόστους ώστε να συμβαδίζει περισσότερο με τα εγχώρια ε, επίπεδα, αυτό, αυτή η φιλοδοξία εντάσσεται στο πρόγραμμα της Επιτροποκρούς ε, και του ψηφιακού προγράμματος της κυρίας Κρούς, το οποίο υποστηρίζουμε πλήρως. Ευχαριστώ, νομίζω ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ θερμά. Έτσι ολοκληρώσαμε αυτήν την γενική συζήτηση και τώρα θα έχουμε μια πιο εντατική συζήτηση για ένα θέμα που ήδη ανέφεραν κάποιοι συνάδελφοι, ε, την πρόταση περιαγωγή 3. Και θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Καράβα από την Κομισιόν, ε, που είναι επικεφαλής ε, της μονάδας, που είναι υπεύθυνη για την πρόταση αυτή για την περιαγωγή. Προτείνω λοιπόν ε, πρώτα ο κύριος Τέραβα να μας παρουσιάσει την πρόταση αυτή και κατόπιν να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μπέρε και ε, να πάρει θέση στο θέμα αυτό. Σας δίνω το λόγο, σας καλωσορίζω θερμά. Παρακαλώ. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Νομίζω ότι είναι πολύ επίκαιρο το θέμα. Είναι πολύ καλή στιγμή να παρουσιάσουμε αναλυτικά την πρότασή μας για το νέο κανονισμό roaming. Όπως ανέφερε ο Κρίς Φοντέιν, η ΠΕΡΕΚ υιοθέτησε χθες, ε, ενέκρινε χθες τη γνωμοδότησή της και νομίζω ότι με τη βάση αυτή θα μπορέσουμε να έχουμε έναν καλό διάλογο για την πρότασή μας. Να δούμε από πού ερχόμαστε και τι μπορούμε να περιμένουμε να συμβεί στην ε, αγορά περιαγωγής εάν υιοθετήσουμε την ε, πρόταση που έχει υποβάλει η Επιτροπή. Πρόθεσή μου με την παρουσίαση αυτή είναι να παρουσιάσω την πρότασή μας με βάση την ε, ανάλυση αδικτύπου που έχουμε κάνει. Να σας παρουσιάσω τα κίνητρά μας για την πρόταση αυτή. Προτού το κάνω αυτό όμως, ε, νομίζω ότι σημαντικό είναι να εξετάσουμε την αγορά περιαγωγής, την κατάσταση στην αγορά και τις ε, ανταγωνιστικές εξελίξεις μέχρι στιγμής. Πρέπει να έχουμε κατά νου το μέγεθος της αγοράς περιαγωγής. Μιλάμε για αγορά 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η περιαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει το 4% των συνολικών εσόδων ε, για, τους, ε, για τις υπηρεσίες κινητών. Και βλέπουμε ότι το 75% των υπηρεσιών αυτών ε, είναι φωνητικές κλήσεις. Τα δεδομένα αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύουν κάτι λιγότερο από 20%. Βλέπουμε όμως ραγδαία αύξηση στον τομέα αυτών. Και νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό μήνυμά μας εδώ, ότι πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι υπηρεσίες περιαγωγής ε, για τη διαβίβαση δεδομένων παίζουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο στις, ε, στην εξέλιξη της αγοράς. Ο παρόν κανονισμός απαιτεί από την Κομισιόν επανεξέταση του κανονισμού περί μέχρι το τέλος ε, του Ιουνίου του 2012 και γι' αυτό ε, έχουμε διεξάγει δημόσια διαβούλευση πέρσι μέχρι τις αρχές της φετινής χρονιάς ε, και έχουμε κάνει ανάλυση αντικτύπου και με βάση αυτή την ανάλυση ετοιμάσαμε την ε, έκθεσή μας ε, σχετικά με την λειτουργία του κανονισμού, την εφαρμογή του κανονισμού και έτσι καταλήξαμε στις 6 Ιουλίου φέτος στις νέες μας προτάσεις. Ποια είναι λοιπόν η κατάσταση στην αγορά περιαγωγής. Εάν κοιτάξουμε τον κανονισμό και την εφαρμογή του, μπορούμε να καταλήξουμε ότι ε, είχαμε καλή συμμόρφωση με τις ε, οροφές των τιμών, με τις ανώτατες τιμές. Ε, οι τιμές έχουν μειωθεί, αλλά παραμένουν στα επίπεδα των ανώτατων ορίων. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι σαφές και ε, συμφωνούν ε, με αυτό ε, νομίζω όλοι οι ενδιαφερόμενοι ότι ο ανταγωνισμός ουσιαστικά δεν είναι αποτελεσματικός και όπως είπε ο Κρίς Φοντέιν σήμερα το πρωί τα διαρθρωτικά προβλήματα στην αγορά περιαγωγής παραμένουν. Ο παρόν κανονισμός λοιπόν έχει ωφελήσει τους καταναλωτές αλλά το διαρθρωτικό πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Αυτό αποτελεί τη βάση για τη νέα μας πρόταση. Εάν κοιτάξουμε ποια είναι η κατάσταση στην ε, αγορά περιαγωγής, όπως βλέπετε από τον πίνακα αυτών, οι τελευταίες μας πληροφορίες ε, δείχνουν ότι οι περισσότεροι πάροχοι υπηρεσιών έχουν τιμές που βρίσκονται κοντά στις ανώτατες ε, τιμές ε, και ότι οι καταναλωτές δεν αποφελούνται από τη μείωση στις τιμές χοντρικής. Λόγω της έλλειψης ανταγωνισμού, οι ε, πάροχοι υπηρεσιών ε, δεν έχουν κίνητρα για να μειώσουν τις τιμές κάτω από τις ε, οριακές τιμές, κάτω από τα ανώτατα, όρια. Αν κοιτάξουμε τις τιμές για τη διαβίβαση δεδομένων, βλέπουμε σε τούτη τη διαφάνεια ότι οι δύο πρώτες στήλες δείχνουν τις τιμές ελληνική και οι δύο τελευταίες μας ε, δείχνουν τις ε, τιμές ε, χοντρικής. Βλέπετε λοιπόν ότι οι τιμές χοντρικής έχουν μειωθεί κατά πολύ και υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις τιμές χοντρικής και τις τιμές λιανικής. Και μάλιστα κατά κάποιο τρόπο σε πολλές περιπτώσεις έχει αυξηθεί το χάσμα. βλέπουμε ότι ε, οι καταναλωτές ε, πληρώνουν ε, πάνω από ένα ευρώ ανά μέγαμπάιτ, ενώ οι χοντρικές τιμές βρίσκονται κάτω από μισό Βασιστήκαμε στα ε, στοιχεία που συνέλεξε η και ε, Έχει συμβάλει σημαντικά στην έκθεση αυτή. Εξετάσαμε λοιπόν το κόστος ε, παροχής υπηρεσιών περιαγωγής. Η ΜΠΕΡΕ έχει κάνει αξιολογήσεις με διάφορες βάσεις, ε, είδε πόσο ε, στοιχίζει μια κλίση ε, με τιμές περιαγωγής, πόσο η αποστολή μηνύματος και πόσο η διαβίβαση δεδομένων. Βλέπουμε ότι οι τιμές αυτές που αντιπροσωπεύουν το κόστος είναι αρκετά χαμηλές σε σχέση με τις τιμές που βλέπουμε στην αγορά αυτή τη στιγμή. για τις φωνητικές κλήσεις ε, οι τιμές ε, κυμαίνονται ανάμεσα σε 5 και 8 ε, λεπτά το λεπτό για, το, για τα μηνύματα ανάμεσα σε 80 cents και 1 με 2 ευρώ και για τα δεδομένα ανάμεσα σε 8 euro cents και 12 ανά Χρειαζόμαστε λοιπόν έναν κανονισμό που θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και αν κοιτάξουμε ποια είναι τα βασικά εμπόδια για τον ανταγωνισμό μπορούμε να τα χωρίσουμε σε τρεις κατηγορίες. Μιλάμε για στρατηγικά, εμπόδια στον ανταγωνισμό, νομοθετικά και διαφορετικά. Η αξιολόγηση αντικτύπου μας επέτρεψε να ε, εξετάσουμε πιο προσεκτικά τις ιδιαιτερότητες ε, της ε, αγοράς περιαγωγής και τα προβλήματα που υπάρχουν στην καρδιά της. Τα προβλήματα που υπάρχουν αφορούν και την ηλιανική και την χονδρική αγορά. Καταρχήν, ε, ένα από τα ε, εμπόδια είναι ότι η περιαγωγή δεν είναι μια ανεξάρτητη υπηρεσία, συνήθως συνδέεται με χώριες υπηρεσίες. Ε, συνήθως ο κατανοτής λαμβάνει ένα πακέτο τιμών, ε, στο οποίο η ένα πακέτο υπηρεσιών, από τα οποία η περιαγωγή αποτελεί μόνο ένα σε ε, επίπεδο χοντρικής, Ο αποκλεισμός ε, των ε, παρόχων υπηρεσιών χοντρικής σημαίνει ότι δεν μπορεί ο πάροχος των λιανικών υπηρεσιών ε, να διαπραγματευτεί άμεσα με ε, τους ε, φορείς σε άλλες χώρες και τέλος η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιο πραγματικό υποκατάστατο των υπηρεσιών περιαγωγής. Υπάρχουν κάποιες τεχνολογίες, μπορεί να αγοράσει κανείς σε μια τοπική αγορά μια τοπική κάρτα ε, κινητού ή να χρησιμοποιήσει το VOIP, ε, αλλά αυτές οι εναλλακτικές λύσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν υποκατάστατο της περιαγωγής, ε, μάλλον μπορούν να θεωρηθούν συμπληρωματικές υπηρεσίες. Οι υπηρεσίε περιαγωγής είναι πολύ εύκολο να χρησιμοποιηθούν. Εάν επιλέξει κανείς μια από τις εναλλακτικέ λύσεις, αυτό αποτελεί επιπλέον προσπάθεια από τον καταναλωτή και γι' αυτό προφανώς οι εναλλακτικέ αυτές λύσεις ε, δεν ε, έχουν επηρεάσει την ε, αγορά υπηρεσιών περιαγωγής και τις τιμές περιαγωγής. Με βάση όλα αυτά λοιπόν υποβάλαμε μία πρόταση η οποία πιστεύουμε ότι είναι υπέρ του ανταγωνισμού. Προτείνουμε να ε, παρατείνουμε το πεδίο εφαρμογής και τη διάρκεια του κανονισμού περιαγωγής μέχρι το 2022. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι σημαντικό. Καθότι εισάγουμε διαρθρωτικά στοιχεία, σημαντικό είναι να υπάρχει νομική και επενδυτική ασφάλεια για τους παράγοντες της αγοράς ώστε να μπορέσουν να υποφεληθούν από τα διαφθορτικά μέτρα που λαμβάνονται. Ε, θεωρούμε λοιπόν υβριδική την προσέγγιση αυτή, διότι παίζουν σημαντικό ρόλο τα διαρθρωτικά στοιχεία, διότι ε, διαβρύνουν την επιλογή του καταναλωτή, ε, ενώ έχουμε κάποια διαθροτικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να παραμείνουν σταθερά ε, σε βάθος χρόνου και επίσης έχουμε ε, κάποιες ε, ανώτατες τιμές που συμπεριλαμβάνουν και τις υπηρεσίες περιαγωγής. Για να κοιτάξουμε πιο προσεκτικά τα διαθροτικά μέτρα που προτείνουμε, θα δούμε ότι Πιστεύουμε ότι θα δώσουν κίνητρα για ε, αύξηση του ανταγωνισμού και ε, όσον αφορά την προσφορά και όσον αφορά τη ζήτηση ε, των υπηρεσιών περιαγωγή. Όσον αφορά την προσφορά, θα είναι πιο εύκολο για εναλλακτικού παρόχου υπηρεσιών να μπουν στην αγορά. Συγκεκριμένα, οι υπάρχοι υπηρεσιών δικτύου θα πρέπει να δώσουν πρόσβαση στα δίκτυα σε άλλου παρόχου υπηρεσιών σε οποιονδήποτε ουσιαστικά ενδιαφέρεται να έχει πρόσβαση στα δίκτυα και να παρέχει υπηρεσίες περιεγωγής. Και ε, η πρόσβαση αυτή θα πρέπει να γίνεται, ε, στη, σύμφωνα, ε, θα πρέπει να γίνεται με τις ρυθμισμένες τιμές χοντρικής που προβλέπονται. Έτσι η εναλλακτική οι πάροχοι υπηρεσιών θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες περιεγωγής. Από την πλευρά της ζήτησης θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και να έχουν περισσότερες επιλογές οι καταναλωτές. Η πρότασή μας... Ε, θα επιτρέπει να υπάρχουν επάροχοι υπηρεσιών ε, για υπηρεσίες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εάν ο καταναλωτής είναι ικανοποιημένος με τον ε, πάροχο υπηρεσιών στη χώρα του, μπορεί να τον κρατήσει για τις εγχώριες υπηρεσίες, αλλά να χρησιμοποιήσει άλλον για τις υπηρεσίες περιαγωγής. Όπως ήδη είπα ταυτόχρονα, θα πρέπει να διασφαλίσουμε την προστασία του καταναλωτή. Θα πρέπει να υπάρχει δίκτυα ασφαλείας για τους καταναλωτές. Είναι σαφές ότι τα διαφορετικά μέτρα θα απαιτήσουν χρόνο για την εφαρμογή τους. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε την σταθερότητα και την προβλεψιμότητα για τους ε, παρόχους υπηρεσιών και να διασφαλίσουμε επίσης και την προστασία του καταναλωτή. Ε, προτείνουμε λοιπόν ε, οι ανώτατε τιμέ ηλιανική να παραμείνουν μέχρι το 2016. Μέχρι τότε το αργότερο περιμένουμε ότι τα διερθωτικά μέτρα θα έχουν αυξήσει τον ανταγωνισμό ώστε να υπάρχουν καινοτόμε πανευρωπαϊκέ προσφορέ ε, υπηρεσιών περιαγωγή, ώστε να μπορούμε να καταργήσουμε τι ανώτατε τιμέ. Εάν όμω αυτό δεν συμβεί, Προτείνουμε πλήρη αναθεώρηση το 2015 που στόχο θα έχει την αξιολόγηση της ε, κατάστασης του ανταγωνισμού στην αγορά καθώς ε, και του επίπεδου των τιμών. Και εάν τότε δούμε ότι η Κομισιόν ήταν υπερβολικά αισιόδοξη, θα υπάρχει ευκαιρία ε, λήψης κατάλληλων μέτρων. Ακούσαμε κάποιες επικρίσεις και νομίζω ότι ο κύριος Φοντέιν θα το αναφέρει αυτό στην απάντησή του στην πρότασή μας. Ε, ακούσαμε κάποιες επικρίσεις σχετικά με την αναθεώρηση του 2015. Ακούσαμε ότι είναι πολύ νωρίς για να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα των διαφορετικών μέτρων που προτείνουμε. Αυτό βέβαια θα αποτελεί σε αντικείμενο συζήτηση στους επόμενους μήνες. Ε, θα ήθελα όμως να τονίσω ότι αν τα διαφορετικά μέτρα που προτείνουμε αποτελούν αξιόπιστη οδό, τότε η αγορά κανονικά θα πρέπει να αντιδράσει σε αυτό από νωρίς. Εάν λοιπόν λειτουργήσει έτσι η αγορά, κανονικά θα δούμε αλλαγές στην αγορά ήδη μέχρι το 2015. Και θα μπορούσε κανείς λοιπόν να υποστηρίξει ότι το 2015 δεν είναι πολύ νωρίς για να γίνει η αξιολόγηση αυτή. Όσον αφορά την ε, διαβίβαση δεδομένων στην περιαγωγή. Είδαμε ότι υπάρχουν ε, παράλογα μεγάλα χάσματα ε, ανάμεσα στις τιμές χοντρικής και λιανικής. Και γι' αυτό προτείνουμε ε, διεύρυνση των ανώτατων τιμών ώστε να καλύπτουν και τις υπηρεσίες δεδομένων μέχρι να ε, τεθεί σε εφαρμογή η διαρθρωτική λύση. Και εδώ προτείνουμε Ε, μέγιστη τιμή ε, για τον καταναλωτή το 2014 ε, μισό ευρώ ανά μεγαμπάιτ. Όσον αφορά την αξιολόγηση αντικτύπου εξετάσαμε διάφορες λύσεις όσον αφορά την ποιότητα, όσον αφορά τον οικονομικό αντίκτυπο και κοινωνικό αντίκτυπο. και έχουμε υπολογίσει επίσης και το κόστος εφαρμογής για τις λύσεις που προτείνουμε. Όπως σας είπα, είχαμε ένα πλήρη κατάλογο λύσεων να διατηρήσουμε την ε, παρούσα προσέγγιση, να ε, καταργήσουμε τη ρύθμιση, να προσαρμόσουμε τις τιμές και κατόπιν εξετάζουμε τα διαρθρωτικά μέτρα, ε, όπως είναι η ξεχωριστή πώληση υπηρεσιών ε, περιαγωγής ε, και τις προσεγγίσεις που βασίζονται στην πρόσβαση στα δίκτυα. Θα επικεντρωθώ στις τρεις λύσεις στις οποίες επικεντρωθήκαμε στην αξιολόγηση αντικτύπου. Η πρώτη λύση είναι να διατηρηθούν ε, οι παρούσες ανώτατες τιμές. Αυτήν την ε, λύση τη διατηρήσαμε για να έχουμε ε, κάποιο μέτρο σύγκρισης. Συγκρίνουμε λοιπόν με τις παρούσες ανώτατες τιμές τις άλλες λύσεις. Η δεύτερη ε, λύση είναι προσαρμοσμένες χαμηλότερες ανώτατες τιμές. Μιλάμε για εισαγωγή ρύθμιση των τιμών. Πρόταση δηλαδή τιμών που να βρίσκονται πολύ κοντά στο ε, κόστος που υπολογίζουμε και ε, τέλος, να έχουμε διαρθρωτικά μέτρα και ε, κάποια σανότετες ε, τιμές για λόγους ασφαλείας. Αν δει κανείς πως έχουν τώρα τα πράγματα, διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταφορά των μειώσεων στην τιμή στη λιανική. Και δεν υπάρχει και ο συντονισμός που απαιτείται γι' αυτό. Αν θέλουμε να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε καλύτερα τις τιμές, Αυτό είναι κάτι το οποίο θα ωφελήσει φυσικά όλους τους τελικούς χρήστες από τις χαμηλότερες τιμές, τους καταναλωτές, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτό θα έχει μόνο προσωρινή δράση, γιατί δεν θα βελτιώσει τον ανταγωνισμό και δεν θα αλλάξει και την δομή της αγοράς. Και δεν ξέρουμε αν θα είναι και συμβατή μια τέτοια ρύθμιση με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου η οποία λέγει ότι ο κανονισμός για την περιαγωγή έχει με τη σωστή νομική βάση αλλά η ρύθμιση των τιμών είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι βασικά προσωρινής φύσης. Και σχετικά τώρα με τα διαφορετικά μέτρα In the και ε, τιμές εγγυήσεων. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διασφαλίσει τον ανταγωνισμό στο μέλλον, χωρίς περισσότερες παρεμβάσεις ε, των ρυθμιστικών αρχών. Προτείνουμε λοιπόν δύο περαιτέρω μέτρα. Καταρχάς ε, τη δυνατότητα πρόσβασης στη χονδρική αγορά, να υπάρξει μεγαλύτερη επιλογή, περισσότερος ανταγωνισμός από εναλλακτικού παροχής και στα πλαίσια συμφωνιών χονδρικής με ξένες εταιρείες, ε, δικτύων και φασμάτων ή και επίσης ε, με επαναγορές συμφωνιών με προηγούμενους, ε, με προηγούμενους παροχής. Και αυτό νομίζουμε ότι μπορεί να οδηγήσει σε πανευρωπαϊκούς παροχής περιαγωγής. Σχετικά απελευθέρωση τώρα των δικτύων, γιατί είναι χρήσιμο κάτι τέτοιο. Πιστεύουμε ότι τα διαφορετικά μέτρα όπως το unbundling είναι βασικό τμήμα της συνολικής λύσης. Η πρόσβαση στη χονδρική από μόνο θα καταστήσει την είσοδο στην αγορά πάρα πολύ δύσκολη. Πρέπει να παρέχουμε στον χρήστη την δυνατότητα να επιλέγει έναν εναλλακτικό χρήστη για τις περιαγωγές του μόνο. Αυτό θα αυξήσει την συνειδητοποίηση του καταναλωτή όπως επίσης και τη διαφάνεια. Γιατί κάτι τέτοιο θα λειτουργήσει σωστά. Ακούσαμε ότι ο κόσμος, ε, οι χρήστες ε, δεν θα συνεχίσουν να συγκρίνουν τις τιμές. Είναι πολύ εύκολο για αυτούς να έχουν τον ίδιο παροχέα για όλες τις ε, υπηρεσίες. Γιατί να αναγκάζεται να κυνηγάει δεξιά και αριστερά τις πιο ενδιαφέρουσες τιμές. Νομίζω ότι η αυξανόμενη ζήτηση για την μεταφορά δεδομένων στα πλαίσια της περιαγωγής μπορεί να οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη ελαστικότητα των υπηρεσιών αυτών και μιλάμε για μια ελαστικότητα πολύ υψηλότερη για τα δεδομένα από ότι για τη φωνητική τηλεφωνία και την τηλεφωνία των μηνυμάτων. Πιστεύουμε λοιπόν ότι οι καταναλωτές είναι όλο ένα και πιο ευαίσθητοι στις τιμές της περιαγωγής και αν τους δίδονται διαφανείς πληροφορίες και αν υπάρχει δυνατότητα εύκολης αλλαγής χρηστών, <coughs> αυτό θα βελτιώσει γενικά τον ανταγωνισμό στις αγορές. Και όπως σας είπα, αυτό θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να είναι εύκολο για τον τελικό χρήστη να κάνει τις αλλαγές που απαιτούνται. Η πρότασή μας λοιπόν είναι να υπάρξει ένας εναλλακτικός παροχέας για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιαγωγή να μπορεί να κρατά βέβαια για να τον χρησιμοποιήσει ο χρήστης τον ίδιο τηλεφωνικό αριθμό, την ίδια κάρτα SIM που χρησιμοποιεί επίσης και για τις τοπικές ε, υπηρεσίες και θα πρέπει να υπάρχει επίσης η δυνατότητα να αλλάζει ανάμεσα στους χρήστες. Να υπογραμμίσω επίσης ότι η πρόταση του κανονισμού είναι τεχνικά ουδέτερη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόσουμε την πρόταση αυτή. Εμείς έχουμε πει στην πρότασή μας, είναι μια πρόταση λεγόμενη διπλή ύμση, double ύμση. Υπάρχουν όμως και άλλες εναλλακτικές λύσεις οι οποίες θα πρέπει να εξεταστούν και να δούμε αν πράγματι μας δίνουν την δυνατότητα για καλύτερο ανταγωνισμό στην αγορά της περιαγωγής. Είπαμε τώρα τις ε, τιμές εγγυήσεων, τις ανώτατες τιμές εγγυήσεων, τις χρειαζόμαστε για τις μεταβατικές περιόδους όπου κάνουμε προτάσεις διαφορετικές και απαιτείται χρόνος για την εφαρμογή τους. Εδώ θα ήθελα να πω ότι αυτές οι ανώτατες τιμές είναι στην ουσία ένα δίκτυο ασφαλείας οι καταναλωτές το 2015-2016 θα πρέπει να μπορούν να ωφεληθούν από τιμές οι οποίες θα είναι χαμηλότερες αυτών που εμείς ονομάζουμε τιμές εγγυήσεων σήμερα. Τώρα για τις οικονομικές επιπτώσεις αυτών των μεθόδων. Εμείς ε, ε, είδαμε ακριβώς τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν αυτά τα οικονομικά μοντέλα τα οποία προτείνουμε. Προσπαθήσαμε να δούμε τις επιπτώσεις αυτών των, προτάσεων και σε σχέση με την ποσότητα των όγκο χρήσης της περιαγωγής και των εισοδημάτων και του κόστου στον καταναλωτή. Αν δει κανεί τις τρεις επιλογές αναλυτικότερα και συγκρίνει λίγο με το υπάρχον αυτή τη στιγμή καθεστώς, διαπιστώνει ότι οι ανώτατες τιμές οι οποίες θα ρυθμίζουν τις τιμές σε επίπεδο κόστους ή πολύ κοντά σε επίπεδο κόστους, προφανώς θα έχουν τις καλύτερες κοινωνικές επιπτώσεις βαχυπρόθεσμα. Θα πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι αυτή δεν είναι μια μακροπρόθεσμη λύση και η τρίτη λύση είναι μια λύση που περιλαμβάνει και το unbundling και την ελεύθερη πρόσβαση και τις ανώτατες τιμές θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας εδώ ότι οι επιπτώσεις αυτές υπολογίζονται επί τη βάση των τιμών ασφαλείας τις οποίες προτείνουμε και ελπίζουμε ότι στο μέλλον οι τιμές θα είναι ακόμα χαμηλότερες, κάτι το οποίο θα βελτιώσει τις δυνατότητες του καταναλωτή και θα δικαιώσει θα έλεγα και την πρότασή μας. Αν εξετάσει κανείς το κόστος εφαρμογής του unbundling βλέπει ότι οι υπολογισμοί οι οποίοι κάνουμε οφείλονται στην τεχνική λύση της διπλής ύμση. Όπως σας είπα, εμείς είμαστε ανοιχτοί και σε άλλες λύσεις, αλλά θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι φιλικές οι λύσεις αυτές και για τον καταναλωτή και ε, ε, θα έλεγα συμβατές επίσης ε, με τον ανταγωνισμό. Το κόστος πάντως των προτάσεων μας θα είναι γύρω στα 300 εκατομμύρια ευρώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λιγότερο από 10% των εισοδημάτων των ετησίων από την περιαγωγή και λιγότερο από 0,2% από, τις, από τα συνολικά έσοδα της, ε, ε, της ασύρματης τηλεφωνίας γενικότερα. Νομίζω ότι στην ουσία εμείς θα δημιουργήσουμε τη βάση για μια υφόρο μορφή ανάπτυξης ε, και ανταγωνισμού στο μέλλον. Πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη λύση, είναι μια επένδυση η οποία αξίζει να γίνει, έτσι ώστε η αγορά της παραγωγής να γίνει πιο ανταγωνιστική και θα καταστήσει τον ανταγωνισμό επίσης πιο ανταγωνιστικό, τον ανταγωνισμό πιο ε, θεμητό και πιο αηφόρο. Πιστεύουμε ότι τα διαφορετικά αυτά μέτρα δίνουν την δυνατότητα καλύτερου ανταγωνισμού στις υπηρεσίες περιαγωγής, μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής στους χρήστες και μακροπρόθεσμα θα δημιουργήσουν ένα πιο σταθερό περιβαλλον ρυθμιστικό. Ε, νομίζουμε ότι θα βελτιωθεί γενικά η, η, λειτουργία της περιαγωγής για τον χρήστη. Κλείνοντας θα ήθελα να πω μετά από μια μακρά σχετικά παρουσίαση ότι η αγορά περιαγωγής δεν λειτουργεί σωστά. Η, η αντιμετώπιση την οποία εφαρμόζουμε από το 2007 για τις ανώτατες τιμές βοηθά τους καταναλωτές αλλά δεν λύνει τα προβλήματα ανταγωνισμού στην αγορά περιαγωγής. Συνεπώς απαιτούνται νέες προτάσεις, απαιτούνται νέες λύσεις οι οποίες θα αντιμετωπίσουν το διαφορετικό πρόβλημα της περιαγωγής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ θερμά για την ε, πολύ πλήρη παρουσίασή σας. Να δώσω τώρα τον λόγο στον κύριο Φοντέιν για να μας παρουσιάσει τις θέσεις του σε σχέση με την πρότασή σας. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη, γιατί όπως είπα στον πρόεδρο πρέπει να φύγω λίγο πριν τις 11.30, αλλά είναι μαζί μου ο κύριος Σίμλετ, που είναι ε, ο επικεφαλής του σχεδίου για την τελική γνωμοδότηση, οπότε είναι σε θέση να απαντήσει σε λεπτομερείς ερωτήσεις. Πρόκειται για μια συνεχιζόμενη διαδικασία που δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί σύντομα. Θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησα στην προηγούμενη μου εισαγωγή, ότι είμαστε πλήρως ε, ε, προσιλωμένοι στο στόχο στήριξης των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Σίγουρα ε, τη στήριξη της Επιτροπής, αλλά και του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου στην επόμενη περίοδο των διαπραγματεύσεων. Μέχρι στιγμής, μέχρι χθε δηλαδή, αυτό που κάναμε είναι ότι από πέρυσι το Δεκέμβριο έχουμε δημοσιεύσει τη γνωμοδότησή μας προς την Επιτροπή για το μέλλον του κανονισμού περιαγωγής, και μάλιστα προσθέσαμε και κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες στην απάντησή μας που δώσαμε το Φεβρουάριο στις διαβουλεύσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχουμε καταλήξει και σε μια τεχνική ανάλυση της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ελπίζουμε ότι έτσι θα διευκρινιστούν πολλά ζητήματα που θα εξεταστούν στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις. Χθες μάλιστα στην ιστοσελίδα μας δημοσιεύσαμε τη σχετική ανάλυση. Θα ήθελα σήμερα να επικεντρωθώ στα θεμελιώδη στοιχεία της ανάλυσης της πρότασής μας. Επίσης θα ήθελα να σχολιάσω και τις μελλοντικές εξελίξεις ε, της αγοράς κινητών για την περίοδο που προτείνει ο κανονισμός που είναι μια μακροχρόνια περίοδος γιατί εκτείνεται μέχρι το 2022 και μιλούμε για μια πολύ δυναμική αγορά. Για να δούμε ποιο θα είναι το όραμά μας ε, στην επόμενη δεκαετία για την περιαγωγή. Καταρχήν μια σύντομη ανάλυση της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε πολλά κοινά στοιχεία αλλά και κάποιες Διαφορέ στην προσέγγιση. Συμφωνούμε φυσικά με το στόχο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μειώσει τι τιμέ, να αυξήσει την διαφάνεια και να ενισχύσει, να διευκολύνει έναν βιώσιμο ανταγωνισμό. Συμπίπτουν λοιπόν οι στόχοι μα. Θεωρούμε όμω ότι τελευταία πέντε ετία ο κανονισμό για την περιαγωγή όντω ωφέλησε σημαντικά του καταναλωτέ. Έχουμε παρατηρήσει μια μείωση των τιμών και ιδιαίτερα προστασία από το σοκ τη λιμπητερή. Βέβαια το κόστος ταυτόχρονα βιώθηκε με γοργούς ρυθμούς. Η διαφορά μεταξύ κόστος και τιμών αυτή τη στιγμή στην αγορά εξακολουθεί να είναι μεγάλη, κάτι που δεν συνάδει με την εσωτερική αγορά. Εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών μελών. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητος εδώ και καιρό αυτός ο κανονισμό. και όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούμε ότι από μόνε τους οι δυνάμει αγοράς δεν είναι αρκετά ισχυρέ για να εξασφαλίσουν λογικές τιμέ για τον καταναλωτή στο εγγύ μέλλον. Χρειαζόμαστε λοιπόν κανονισμό και χονδρική και ελληνικής και φυσικά ανώτατα όρια λιανικής. Συμφωνούμε επίσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι οροφές τιμών θα πρέπει να μειώνονται σταδιακά για να πλησιάσουν το κόστος, γιατί εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική διαφορά χάσμα μεταξύ τιμών και κόστους και να προσαρμοστούν σε αντίστοιχε ισοδύναμε τιμέ τη εσωτερική αγορά. Αυτό είναι ο στόχο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε οι τιμέ περιαγωγή μέχρι το 2015 να πλησιάσουν στι ε, τοπικέ τιμέ, σε χώρε τιμέ περιαγωγή. Τώρα, μέσω πρόθεσμα, οι μειώσει ε, του κόστου χονδρικής θα πρέπει να δώσει την ευκαιρία στους φορείς εκμετάλλευση να προσφέρουν ε, στους πελάτες τους ένα ενιαίο ευρωπαϊκό τιμολόγιο και οι πελάτες να πληρώνουν για ανταλλαγή μηνυμάτων ε, κλήσεις με λογικές τιμές. Φυσικά ακόμη έχουμε μεγάλη απόσταση από αυτό το στόχο, αλλά θα σημειώσουμε πρόοδο με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, για την περιαγωγή δεδομένων. Καλωσορίζουμε την πρόταση για νέε τιμέ εξασφάλιση, ανώτερε τιμέ ό,τι αφορά την περιαγωγή δεδομένων. Λιανική, μάλιστα. Και μάλιστα ε, έχουμε στην αγορά αρκετά ελκυστικά προϊόντα και τιμές, αλλά δυστυχώς δεν είναι παντού προσιτές στην Ένωση και πολλές τιμές στην Ένωση εξακολουθούν να είναι αδικαιολόγητα υπέρογες. Οι, οι οροφές των τιμών θα πρέπει να απαλείψουν τις υπέρογες τιμές που χρεώνονται ακόμη και σήμερα σε πολλούς για την περιαγωγή δεδομένων. Θα πρέπει να γίνει κάποια εξισορρόπηση, αλλά αυτή η εξισορρόπηση φυσικά θα πρέπει να παραβλάψει τον ανταγωνισμό της ε, περιαγωγής δεδομένων. Βέβαια έχουμε και εναλλακτικέ λύσεις όπως το Wi-Fi που ασκούν ανταγωνιστικές πιέσεις στην αγορά. Παρ' όλα αυτά ε, αξίζει να τονίσουμε ότι οι ανώτερες τιμές ελάχιστα θα ευνοήσουν τους ε, μεγάλους χρήστες τους, ε, της Έχουμε όλο και περισσότερους χρήστες smartphones. Βέβαια χρειαζόμαστε μικρότερες τιμές ώστε ε, να μπορούν να χρησιμοποιούν με λογικές τιμές και τα smartphone. Να αποφύγουμε παράδοξες καταστάσεις βέβαια. Με, στο μέσο που η ζήτηση αυξάνεται θα μειωθούν οι τιμές. Οπότε έχουμε ε, ελπίδες ότι στο μέλλον θα βελτιωθεί η κατάσταση. Φυσικά θα εξακολουθούμε να παρακολουθούμε τις εξελίσεις. Ό,τι αφορά τις ε, διαρθρωτικές λύσεις. Κανένας δεν θέλει μια τέρμονη ρύθμιση τιμών. Ούτε και ο Μπερέκ. Συμφωνούμε λοιπόν ότι παράλληλα με τα ανώτατα όρια και τις ε, ασφαλιστικές δικλείδε θα πρέπει να βρεθεί και μια διαρθρωτική λύση. Μια διαρθρωτική λύση που θα διορθώνει τις αδυναμίες αγοράς, θα ενισχύει τον ανταγωνισμό μέχρι ότου αφαιρεθεί, εξαλειφθεί αυτή η ρύθμιση των τιμών. Χρειαζόμαστε μια λύση ε, που θα είναι ταχεία και εύκολη εφαρμογή. Αλλιώ θα χάσουμε το παράθυρο τη ευκαιρία και πολύ πιθανό οι εξελίξεις ε, της αγοράς να προσφέρουν λύσεις, αλλά χρειαζόμαστε γοργές λύσεις. Επίση, ε, χαμηλότερα, χαμηλότερο κόστος περιαγωγής θα διευκολύνουν μια πανευρωπαϊκή λύση και δεν αξίζει μια λύση που θα είναι ε, δαπανηρή σε ό,τι αφορά τα, τα ωφέλη που περιμέναμε από αυτήν. Ο Μπερέκ πιστεύει ότι μία απόλυτα ικανοποιητική διαρθρωτική λύση δεν έχει προταθεί και όταν εννοώ ικανοποιητική λύση, εννοώ μια λύση που θα εξασφαλίζει τον ανταγωνισμό και ωφέλη στους καταναλωτές που θα είναι ανάλογα προς την ε, ε, εμπορική και τακτική εφαρμογή. Προς... Προτείναμε κάποιες πρακτικές λύσεις ε, το Δεκέμβριο και το Φεβρουάριο, γιατί δεν μας ικανοποίησαν οι προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ό,τι αφορά τον έλεγχο επιπτώ... τη μελέτη επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε ό,τι αφορά την ε, χωριστή χρέωση για τη διεθνή ταυτότητα, διπλή διεθνή ταυτότητα κινητού η IMCI. Έχουμε κάποιες επιφυλάξεις, παρόλο που θεωρούμε ελκυστική αυτή την πρόταση. Έχουμε αφιβολίες για τα ωφέλη. Κάποια άλλα μέτρα χρονικής που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μείωση των τιμοχονδρικής, μαζί με μια γενική πρόσβαση χονδρικής, πιστεύουμε ότι θα εξασφαλίσουν ε, και μεσοπρόθεσμα ωφέλη στον ανταγωνισμό. Και κάτι τέτοιο ίσως ε, επιτρέψει σε φορείς εκμετάλλευσης τη δυνατότητα να προσφέρουν πιο ε, ελκυστικές τιμές περιαγωγής, ιδιαίτερα σε μελλοντικά πακέτα. Επίσης θα διευκολύνουν την ε, εισαγωγή νέων ε, φορέων στην αγορά με το στόχο μιας οικουμενικής υπηρεσίας SIM, διαχείριση συνδρομητικών πληροφοριών. Υπάρχει κίνδυνος αυτή η διπλή λύση MCI να δώσει ελάχιστα επιπλέον ωφέλη. Προτιμούμε τα άλλα μέτρα της χονδρικής. Πάντως πιστεύουμε ότι οι λύσεις αυτές θα συνδυαστούν με κάποια εφαρμοστικά μέτρα και με συνεχείς μελέτες. Και το ζητούμενο φυσικά είναι μια αγοργή εφαρμογή, γιατί θα μειωθούν τα εφέλη αν η εφαρμογή είναι αργή. Βέβαια έχουμε όλο και νέες ε, ε, εναλλακτικέ λύσει για την αποδέσμευση, αποδεσμοποίηση, αλλά δεν μπορούμε να επιλέξουμε ακόμα. Είναι πολύ για να δώσουμε έμφαση σε μία λύση. Θέλουμε από κοινού με τη βιομηχανία να εξετάσουμε και να αναλύσουμε τις διάφορες αναλεκτικές αναζητώντας το συντομότερο δυνατό την κατάλληλη λύση. Πάντως, ε, στο έγγραφό μας ε, απευθύνουμε κλίση στην Επιτροπή να λάβει απόφαση προκειμένου να επιλέξει συγκεκριμένη διαρθρωτική λύση που θα πρέπει να επιλεγεί μόνο εφόσον εξασφαλιστεί η παροχή ωφελών σε όλους τους καταναλωτές και τους ε, συστηματικούς χρήστες αλλά και τους περιστασιακούς. Επίσης θα πρέπει αυτή η λύση να εφαρμόσει σχετικά γρήγορα και με οικονομικό τρόπο, να μην είναι υπερβολικά δαπανηρή. Επίσης χρειαζόμαστε μια κρίσιμη μάζα ε, φορέων της αγοράς. Και φυσικά θα, θα πρέπει να ενισχύει τον ανταγωνισμό. σε περίπτωση που δεν έχουν εμπορικά ωφέλη φυσικά, οι φορεί δεν πρόκειται να εφαρμόσουν κάποιε τέτοιε λύσει. Πάντω, είμαστε ανοιχτοί στι συζητήσει και συνεργαζόμαστε με τη βιομηχανία και την Επιτροπή προκειμένου να ε, καθορίσουμε κάποιε κατευθυντήριε γραμμέ για να υποστηρίξουμε την εφαρμογή. Αυτό και έχουμε κάπως πιο επιφυλακτική λύση ως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα, τα αποτελέσματα των διαρθρωτικών ε, λύσεων. Φυσικά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ε, εύρυθμη λειτουργία της αγοράς πριν απαλείψουμε, τη ρυθμίση των τιμών. Φυσικά μερικοί ζήτησαν ε, τα χάσματα, οι διαφορές τιμών να απαλληφθούν το συντομότερο δυνατόν. Συμφωνούμε, αλλά ακόμη είναι πρόημο να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος και δεν θα πρέπει να διακινδυνεύσουμε την προστασία του καταναλωτή. Και φυσικά, αν τα επόμενα χρόνια παραμείνουν αυτές οι ανώτατες τιμές ε, ελληνικής, θα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το ύψος τους. Αυτό είναι πολύ επιμαχό θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θέλει να ενισχύσει τον ανταγωνισμό και από αυτή την άποψη δεν θα ήταν σκόπιμο να έχουμε χαμηλά, τόσο χαμηλά ανώτατα όρια που θα αποτρέπουν ε, νέους ε, φορεί από την εισαγωγή στην αγορά. Ούτε θα πρέπει να είναι πολύ ψηλά, ψηλά αυτά τα ανώτατα όρια, ώστε να μην εξασφαλίζουν μείωση των τιμών. Θα πρέπει εδώ να βρούμε μια σωστή ισορροπία. Πάντως, αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Μπερέκ πάντως θα έδινε μια διαφορετική αντίληψη αυτής της ισορροπίας. Προτείνουμε από το 2014 κάποιες χαμηλότερες ανώτερες τιμές. Πιστεύουμε ότι ένα περιθώριο 200% ε, λιανικής, που είναι τριπλάσιο της ε, χονδρικής ε, ε, που πληρώνουν οι φορείς πιστεύουμε ότι αρκεί για να εξασφαλίσει είσοδο νέων φορέων αλλά και να εξασφαλίσει μια αποτελεσματικότητα του ανταγωνισμού. Γιατί όσο ενισχύεται ο ανταγωνισμό, τόσο θα εξασφαλίσει και η προστασία του καταναλωτή. Δεδομένων των ε, αβεβαιοτήτων και του μακροχρόνιου χρονικού ορίζοντα του κανονισμού, ο Μπερέκ πιστεύει ότι η αναθεώρηση του 2015 θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ξενυχιστική μεταρρύθμιση της στρατηγικής. Γιατί η αγορά είναι πολύ δυναμική και ήδη και μια τριετή είναι μεγάλη. Θα πρέπει επίσης να γίνει μια επαναθεώρηση του κατά πόσο η ε, δυνάμει αγορά, ε, άσχετα από το κατά πόσο ενισχύθηκαν από τα διαρθρωτικά μέτρα, όντω έχουν μια επιρροή στη διαμόρφωση των τιμών. Επίση θα πρέπει να αναλύσουμε κατά πόσο οι προσδοκίε που έχουμε για το κόστος για την επόμενη δεκαετία έχουν υλοποιηθεί. Η δεκαετία είναι ε, πολύ μεγάλο διάστημα για να ορίσουμε ρυθμιστικέ ανώτατε τιμέ σε ένα τόσο δυναμικό περιβάλλον όπω είναι αυτό τη κινητή ε, τηλεφωνία. Εμείς κάθε διετία ή τριετία έχουμε τέτοιες ε, αναθεωρήσεις στα πλαίσια του πλαίσιου, ακριβώ λόγω του δυναμικού χαρακτήρα αυτής της αγοράς. Τέλος, η ανάλυση, η αναθεώρηση, η εκτίμηση θα πρέπει να δείξει κατά πόσο χρειάζομαστε, εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε τέτοιες ανώτερες τιμές, ποια θα πρέπει να είναι τα επίπεδά τους και οι διαφορές τους από τις τιμές ελληνικής. Διαφορά δηλαδή του επίπεδου χονδρικής από το επίπεδο λιανικής. Τέλος, ε, θα ήθελα να αναφέρω κάτι που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμά μας και που όμως δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Μπερέκ θα ήθελε να συμπεριληφθεί αυτό το θέμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ αποτελεσματικούς μηχανισμούς προστασίας από το σοκ του λογαριασμού που ξεκίνησε το 2010 και κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να επεκταθούν και να εφαρμόζονται και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζουμε βέβαια ότι ήταν δύσκολη εφαρμογή αρχικά οι κανόνες, αλλά τελικά έχουμε α, γλιτώσει τα σενάρια τρόμου καταναλωτών που επιστρέφουν από τις διακοπές και αντιμετωπίζουν αστρονομικά τιμολόγια. Τέτοιες ιστορίες δεν έχουμε εντός της Ευρώπης, αλλά δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν εκτός Ευρώπης και κάποιοι φορείς εκμετάλλευσης και ο θελό έχουν εισαγάγει κάποια μέτρα που όμως ε, είναι ανεπαρκή κατά τη γνώμη του Μπερέκ. Πιστεύουμε ότι μια τέτοια διεύρυνση των μέτρων θα μπορούσε να είναι εύκολη εφαρμογή και σχετικά φθηνή. Να ισχύει και για του ε, καταναλωτέ που ταξιδεύουν εκτό Ευρώπη και δικαιολογείται και ω μέτρο εσωτερική αγορά. Γιατί η λιανική ε, περιαγωγή δεδομένων γίνεται από εταιρείε, γίνεται του άλλου από εταιρείε εντό τη Ένωση για καταναλωτές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν κατακλείδη, η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πιστεύουμε ότι είναι θεμελιώδη σημασία ε, να προασπίσουμε τα συμφέροντα όλων των καταναλωτών. Έχουμε κάποιε προτάσει που πιστεύουμε ότι θα ενισχύσουν την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είμαστε υπέρ της διαμόρφωσης μιας διαρθρωτικής λύσης, μιας λύσης όμως που θα ενισχύει τον ε, ανταγωνισμό στην διεθνή αγορά περιαγωγής, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Βιομηχανία και αν συμφωνείτε από κοινού και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ως προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελα να πω ότι είμαστε στη διάθεσή σας για τεχνική υποστήριξη προκειμένου να διαμορφώσετε μια πιο τεκμηριωμένη γνώμη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας αυτή. Ε, μας παρουσιάσατε τη θέση σας ε, σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν. Μια σειρά συναντέρφων ζήτησαν το λόγο. Ε, με τη σειρά, ας τους πάρουμε, η κυρία Δελκαστήγιο. Εν συντομία, για να προλάβει να μ' ακούσει και ο κύριος Φοντέιν πριν φύγει ευχαριστώ θερμά για την ε, ανάλυση αντικτύπου που έκανε ο ο Φορέας ε, των Ρυθμιστικών Αρχών. Γιατί η γνωμοδότηση του Μπερέκ είναι απαραίτητη στην περίπτωση αυτή. Είναι αναφίβολο ότι ο στόχος μας είναι κοινό. Θέλουμε μια πιο ανταγωνιστική αγορά και επίσης μια ολοκληρωμένη αγορά και για την κινητή τηλεφωνία και για, τα, για τις κλήσεις και για, τη, για τα μηνύματα και για τα δεδομένα. Εγώ χθε σε συντομία έριξα μια ματιά στην έκθεση του Μπερέκ και σήμερα με την εισαγωγή συμπληρώθηκε η εντύπωση που σχημάτισα. Οπότε τα σχόλιά μου έχουν το χαρακτήρα του brainstorming. Δεν είναι αποκρισταλωμένες απόψε, καμία περίπτωση, γιατί εντός ολίγου θα ξεκινήσει η διαδικασία στο Συμβούλιο και θα εμβαθύνουμε στο θέμα αυτό. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον να χρησιμοποιήσουμε ως αφετηρία την έκθεση του Μπερέκ. Διαβάζοντας την έκθεση και ακούγοντας την παρουσίαση του Διευθυντού, και χωρίς να γνωρίζει την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι είναι ελάχιστε οι διαφορές και η διαφορά μεταξύ πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ανάλυση του Μπερέκ θα μπορούσε να συνοψιστεί ως, ως διαφορά επουσιώδου σημασία, ως διαφορά αποχρώσεων. Αλλά νομίζω ότι η διαφορά είναι πολύ πιο σημαντική, δεν αφορά κάποιες μικρές αποχρώσεις. Και θα ήθελα εδώ να κάνω και λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Ποιο είναι το βασικό επιχείρημα της ανάλυσης του Μπερέκ. Το ότι δεν αρκεί μία διαρθρωτική μεταρρύθμιση, όπως αυτή που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν δεν έχουμε από κοινού με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και κάποια διατήρηση των οροφών των τιμών, των price caps και ε, προτάσεις για, τη, για το wholesale, τη χονδρική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι όταν υποβάλλονται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις δεν χρειάζονται πια οι οροφές στις τιμές. Ενώ ο Μπερέκ λέει ακόμη και αν ξεκινήσουν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις χρειαζόμαστε για ένα βαθμό, για μια περίοδο ακόμη τις οροφές των τιμών, μέχρι ότου μπορέσουμε να αξιολογήσουμε κατά πόσο αυτά τα μέτρα ενισχύουν τον ανταγωνισμό ή τον αναχαιτίζουν. Οπότε θα ήθελα εδώ να επισημάνω δύο θέματα που δεν έχω καταλάβει ακόμη. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αναγνώριση ότι οι φορείς εκμετάλλευσης τήρησαν τις απαιτήσει των κανονισμών 1 και 2. Και από αυτή την άποψη υπάρχει μια εμπιστοσύνη ότι οι φορείς εκμετάλλευσης και έγκαιρα και πιστά θα τηρήσουν τις απαιτήσεις και του νέου κανονισμού και τις προτάσεις για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Όλος παραδόξως υπάρχει μια δυσπιστία από ό,τι φαίνεται του Μπερέκ πολύ μεγαλύτερη από την δυσπιστία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεύτερο πρόβλημα είναι το κόστος, τα κόστη. Γιατί δεν θα είναι καθόλου εύκολο να εφαρμόσουμε εμπράκτο στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Από τεχνική άποψη το θέμα είναι πολύ περίπλοκο. Μπορεί να φαίνεται απλό να αλλάζει κανείς ε, φορέ εκμετάλλευση που ταξιδεύει, αλλά δεν είναι καθόλου απλό. Είναι πολύ σύνθετο ζήτημα και φυσικά θα χρειαστεί και μια ευρηματικότητα και από τεχνική άποψη. Και αν σε αυτό προσθέσουμε την ανάγκη μείωση των ε, ανώτατων ωραρίων, ορίων συγγνώμη, τιμών για τη χονδρική, ερωτώ αν έτσι θα έχουμε αρνητικό αντίκτυπο σε ό,τι αφορά τον αριθμό των φορέων εκμετάλλευσης που μπορούν να μπουν στην αγορά της περιαγωγής. Γιατί αν ο συνδυασμός των επενδύσεων με τη μείωση των ανωτάτων ορίων τιμών στη χονδρική διατηρηθούν, ίσως αποτρέψουν αντί να ενθαρρύνουν νέους φορείς να ενταχθούν στην αγορά του ρόμικ. Δεν έχει αποδειχθεί ο αντίκτυπος ενός τέτοιου συνδυασμού. Αυτές είναι οι πρωταρχικές μου σκέψεις. Και λαμβάνοντας υπόψη το πώς στο παρελθόν ε, λειτουργήσε η νομοθεσία, ο κανονισμός 1 και 2 για την περιαγωγή, πιστεύω ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και ακούσαμε την επιχειρηματολογία. Αλλά αυτό το θέμα θα παραμείνει ανοιχτό και στη συζήτηση του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί ίσως είμαστε το πιο ευαίσθητο κοινοβούλιο του κόσμου σε ό,τι αφορά την ανάγκη εξασφάλισης μιας ανταγωνιστικής αγοράς και για τους ε, πολίτες που μετακινούνται. Γιατί ακριβώς ε, ε, εμείς πληγόμαστε από την έλλειψη μιας ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σε περίπτωση που κανείς ταξιδεύει πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε και νέα επιχειρήματα. Αν ναι, παρακαλώ να τα ακούσουμε. Πάντως, ακόμη και αν δεν έχετε σήμερα, δεν πειράζει, γιατί θα έχουμε πολλές ευκαιρίες και στο μέλλον να ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό με τον Μπερέκ. Ο κύριος Ρουμπίχ. Ευχαριστώ για την καλή μελέτη αυτή και για τις καλές πιστεύω προτάσεις. Πιστεύω ότι πρέπει να ρωτήσω, οι προβλεπόμενες ανώτατες τιμές ε, στην περιαγωγή δεδομένων, όταν κοιτώ σήμερα τη συσκευή μου, βλέπω ότι 100 ε, κιλομπάιτ ε, στοιχίζουν 0,99 ή 1,39 ευρώ. Αυτές είναι οι δύο ανώτατες τιμές και έχουμε εμείς ταξιδεύουμε συχνά σε όλη την Ευρώπη. Αλλά μήπως θα πρέπει να υπάρχει ένα πρακτικό παράδειγμα. Όταν κανείς κατεβάζει ε, μία ταινία που διαρκεί ε, μία... Ε, διαρκεί μία ώρα, αυτό είναι ένα γιγαμπάιτ. αυτό σημαίνει ότι πληρώνει κανείς 9.900 ε, ε, ευρώ για ένα γίγαμπάιτ ή αντίστοιχα 13.900. Ενώ στην Αυστρία, εάν κατεβάσω ένα γίγαμπάιτ, αυτό μου στοιχίζει ένα ευρώ. Δηλαδή, αν κατεβάσω αυτή την ταινία της μίας ώρας στο σπίτι μου, ε, πληρώνω ένα ευρώ. Εάν ε, αυτό το κάνω σε άλλη χώρη πληρώνω 13.900 ε, ευρώ. Εσείς πώς καταλήγετε στα 500 ευρώ. Ευχαριστώ. Μήπως εξαρτάται από το ποια, ε, περί ποιας πρόκειται. Ε, από αυτό μάλλον θα εξαρτηθεί η απάντηση των ερωτήσεων. Ο συνάδελφος Νίστελ Ρόι. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Άκουσα με προσοχή τις προτάσεις σας. Θα προτιμούσαμε να τις συζητήσουμε αναλυτικότερα στο Στρασβούργο, αλλά εν πάση περιπτώσει έστω και σήμερα δεν είναι κακό. Πήραμε λοιπόν πολλά στοιχεία, πολύ περισσότερα από ό,τι είχαμε την τελευταία φορά ε, στη διάθεσή μας. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να οργανώσουμε μια ακρόαση γύρω από το θέμα αυτό γιατί καλό θα είναι να μπορέσουμε να ζυμώσουμε όλες αυτές τις ιδέες που προέρχονται από τους εμπλεκόμενους, τους ενδιαφερόμενους και να δούμε τι επιπτώσεις από τις προτάσεις αυτές θα υπάρξουν στο μέλλον. Άκουσα προσεκτικά αυτά που είπατε για το τι συμβαίνει στον τομέα της περιαγωγής. Εάν πράγματι θέλετε να κάνετε κάτι το πάρα πολύ ε, σημαντικό, θα πρέπει εσείς να στοχεύσετε τις τιμές φυσικά. θα πρέπει οι τιμές αυτές να έρθουν πολύ κοντά στις λεγόμενες εθνικές τιμές. Στα πλαίσια του υπάρχοντος κώδικα νομίζω ότι τα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις έχουν αυξηθεί. Αυτό είναι λίγο περίεργο με τη μείωση των τιμών. Αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να προσπαθήσετε να δείτε ε, πώς μπορούμε να φτάσουμε στο λεγόμενο εθνικό επίπεδο των τιμών. Υπάρχουν τεχνικές δυνατότητες για την πιθανότητα και την δυνατότητα επιλογής του παροχέα της περιαγωγής. Νομίζω ότι μπορούμε να τα βρούμε αυτά, αλλά αυτά θα πρέπει να τα κάνουν οι τεχνικοί. Το να πούμε ότι το 2022 θα αλλάξουν τα πράγματα είναι πάρα πολύ μακριά. Θα πρέπει να αλλάξουν μέχρι το 2015. Η αίσθησή μου είναι ότι τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται δεν είναι ουσιαστικά, είναι ημίμετρα. Αυτοί οι οποίοι πραγματικά θέλουν να στηρίξουν τον ανταγωνισμό θα το πετύχουν γιατί ε, γνωρίζουν πώς. Μέτσαρος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την ΠΕΡΕΚ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις παρουσιάσεις που έκαναν. Χαίρομαι που το συζητάμε το θέμα αυτό τώρα και θα ήθελα να ζητήσω και την ΜΠΕΡΕΚ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβουν υπόψη τους τις μικρότερες χώρες γιατί οι μικρότερες χώρες ε, δυστυχώς πάντα χάνουν όταν ερχόμαστε να συζητήσουμε τις διαφορές ανάμεσα στις χώρες. Η Ουγγαρία, η Βουλγαρία βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Δεν ξέρω βέβαια τι κατάσταση επικρατεί στην Πολωνία. Υπάρχουν όμως εκεί τεράστιες διαφορές σχετικά με τις τιμές ε, τις οποίες προσφέρουν οι παροχείς. Πολλές φορές ε, η μία τιμή είναι δεκαπλασία της άλλης. Ιδιαίτερα το συγκρίνουμε με το κόστος της ε, κινητής φωνητικής τηλεφωνίας. Ο κύριος Φοντέιν, ο εκπρόσωπος της Μπερέκ, είπε ότι θα χρειαστούν περισσότερες ρυθμίσεις και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Καλό είναι το ότι το λέτε αυτό, καλό είναι που αναφέρεστε και σε ευρωπαϊκά τιμολόγια και ελπίζω κάποια στιγμή να καταλήξουμε στα λεγόμενα ευρωπαϊκά τιμολόγια γιατί αυτό είναι προς όφελος και των μικρομεσαίων, μικρών και μικρομεσαίων παροχέων. Δεν μπορούμε να εξαρτηθούμε απόλυτα και αποκλειστικά στις δυνάμεις της αγοράς. Τα πράγματα είναι αρκετά πιο περίπλοκα. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει το ταχύτερο δυνατόν, σχετικά γρήγορα εν πάση περιπτώσει, γιατί αυτό είναι απαραίτητο για τις λεγόμενες μικρές χώρες. σχετικά τώρα για τα κέρδη άνω του 110%. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς φυσικά δικαιολόγητο. Είναι σαφές ότι θα πρέπει τα ποσοστά αυτά, ιδιαίτερα στις μικρές χώρες, να αλλάξουν. Στη Σλοβακία υπάρχουν τρεις παροχές και δεν ξέρω αν θα υπάρξουν και περισσότεροι στο μέλλον. Μπέρετ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον αυτά που είπε ο κύριος Φοντέιν και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που σχολίασε και όλα στις προτάσεις του κύριου Φοντέιν. Δύο μικρές παρατηρήσεις μόνο, ιδιαίτερα προς τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορείτε μήπως να μας δώσετε μια κάποια ιδέα συγκρίσεων με άλλες αγορές, Ηνωμένε Πολιτείε, Νότια Κορέα. Ποια είναι τα περιθώρια κέρδους για τους παροχείς τελεκόμ είναι στο ίδιο επίπεδο του 110% αλλά προφανώς εμείς θέλουμε να δώσουμε περιθώρια στις επιχειρήσεις μας για να μπορούν να επενδύουν και σε νέες τεχνολογίες. Δεύτερο θέμα, αναφερθήκατε στην ταχεία αύξηση της χρήσης των, της περιαγωγής δεδομένων, είναι το 20% της περιαγωγής σήμερα και αυξάνεται συνεχώς. Όταν η πρόταση αυτή μετατραπεί σε κανονισμό ελπίζουμε ότι η αύξηση αυτή θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ε, αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα σε, ε, ηλεκτρονικό συνοστισμό στην αγορά. Και μπορούμε σε τεχνικό επίπεδο εμείς να ανταποκριθούμε ακριβώς σε αυτόν τον συνοστισμό, στην αυξημένη εν περιπτώσει και θα ακολουθήσουν αυξήσεις και βελτιώσεις στον τομέα των, των επενδύσεων έτσι ώστε να καλυφθούν οι νέες ανάγκες. Εάν συμφωνείτε, θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο... Θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή ώστε να δώσουμε στον κύριο Φοντέιν τη δυνατότητα να απαντήσει σε ερωτήσεις που ήδη τέθηκαν. Δεν είναι δίκαιο αυτό. Καλά, τότε θα προχωρήσουμε. Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη, αλλά και άλλες ομάδες έχουν ερωτήσεις ε, προς τον κύριο Φοντέιν, αλλά δίνετε ε, συνεχώς το λόγο στο ΕΛΚ. Ξέρω ότι είναι η ομάδα σας, αλλά ε, μήπως να, να είσαστε πιο δίκαιος. Εντάξει, θα δώσουμε τότε τη δυνατότητα σε άλλους συναδέλφους να θέσουν ερωτήσεις και κατόπιν θα απαντήσει ο συναδελφός σας. Εντάξει, καταλαβαίνω. Η κυρία Χέρτσογκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, και εγώ ήθελα να αναφέρω ότι πιστεύω ότι η γραμματεία θα πρέπει να ε, πετύχει πιο καλή ισορροπία ε, προς όφελος ε, της ειρήνης στην Επιτροπή μας. Νομίζω ότι είναι καλύτερη ιδέα αυτή. Δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, νομίζω ότι η περιεγωγή ήταν για την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία ένα από τα σημαντικότερα θέματα και είναι ίσως το μόνο θέμα της Επιτροπής μας που τέθηκε στις ευρωεκλογέ. Εμείς λοιπόν ως Κοινοβούλιο νομίζω ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό πριν το 2014 διότι μιλάμε για το ευρωπαϊκό εγχείρημα, μιλάμε για ένα θέμα το οποίο όχι μόνο βοηθάει στην εκλογή των μεμονωμένων πολιτικών ομάδων αλλά αυξάνει και τη συνείδηση των Ευρωπαίων ε, πολιτών ε, για, όσον αφορά την ε, Ευρώπη. Νομίζω ότι μετά από την αλλαγή της νομοθεσίας αυτής, αν μπορούμε να δούμε σημαντικό αρνητικό αποτέλεσμα ε, στο, στη τσάντα του καταναλωτή. Εγώ έχω μόνιμα τρία ή τέσσερα κινητά τηλέφωνα στη τσάντα μου. Ε, αν ε, είναι δυνατό να επιλέγω πάροχο υπηρεσιών, τότε χρειάζομαι μόνο ένα κινητό και θα χρειάζομαι έτσι μικρότερη τσάντα. Αυτή λοιπόν θα είναι η αξία της πρότασης αυτής. Ε, εάν λοιπόν είναι δυνητό κάτι τέτοιο, τότε οι ε, πελάτες, και όχι μόνο οι γυναίκες ε, που κρατάνε σαντούλες, και οι άντρες θα ε, επιλέξουν ε, ε, μονομενα στοιχεία, για παράδειγμα, για το οικογενειακό πακέτο. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω ένα κινητό για την οικογένειά μου, ένα για τα, τα μέλη της ομάδας μου, ένα για το Βέλγιο, ένα για τη χώρα μου κλπ. Εάν όμως είναι δυνατή η επιλογή, θα ήθελα πολύ να έχω ένα κινητό και με, πατώντας ένα κουμπί να επιλέγω τον πάροχο. Εάν λοιπόν είναι σωστό αυτό που οραματίζομαι, τότε με την ε, νομοθεσία αυτή θα έχουμε τη ε, δυνατότητα να αλλάξουμε την ε, αγορά κινητών. Και αν τεχνικά είναι εφικτό αυτό, και ελπίζω να είναι τεχνικά εύκολο να γίνει, τότε θα υπάρχει ο αυξημένος κίνδυνος οι καταναλωτές Ε, να ξεχνιούνται ε, Εάν είναι πολύ εύκολο να γίνει η επιλογή, τότε είναι πολύ εύκολο να ξεχάσει κανείς ε, και έτσι να λαμβάνει υπηρεσίες υπηρεσίε που δεν ήθελε. Όπως ακούσαμε λογαριασμούς χιλίων ευρώ σε μήνα του μέλητος επειδή είχε ξεχάσει ο καταναλωτής να αλλάξει πάροχο. Πώς λοιπόν ε, μπορούμε να φροντίσουμε ε, να μην γίνεται αυτό. Συμφωνώ απόλυτα ότι θα πρέπει να είναι πιο απλοί οι λογαριασμοί και να σας πω ε, τη δική μου εμπειρία έχοντας εξετάσει τους λογαριασμούς μου επί δύο μέρες κατέληξα σε ποιον πάροχο υπηρεσιών ήθελα και τελικά δύο μέρες έμεινα χωρίς ε, κινητό. Δύο μέρες ε, με πήρε μαζί με τον τεχνικό εμπειρογνώμο να καταλήξω στη σωστή λύση. Θα πρέπει λοιπόν να είναι πιο απλές οι επιλογές. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Λάμπερτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα μια ερώτηση προς την Κομισιόν. Όταν κάνατε την πρότασή σας και μετά από τη δημόσια διαβούλευση. Ήρθατε σε επαφή και με τις ενώσεις των καταναλωτών στην Ευρώπη, ιδιαίτερα σε σχέση με τα διαρθρωτικά μέτρα, όχι μόνο τα ανώτατα όρια, γιατί εκεί προφανώς θα συμφωνούν, αλλά πιστεύετε ότι τα διαφθρωτικά μέτρα τα οποία εσείς προτείνετε είναι κατάλληλα για τους καταναλώτες, πώς το κρίνουν αυτοί. Ελπίζω να ήρθατε σε επαφή και να διαβουλευθήκατε και μαζί τους και να πήραν μέρος στην επίσημη διαβούλευση την οποία κάναμε. Δεύτερον, θα ήθελα να μάθω από την Μπερέκ αυτά που είπε για τις ανώτατες τιμές. Συμφωνώ με τις ε, ε, ότι τα ανώτατα όρια για μεγάλα χρονικά διαστήματα δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα πρακτικό. Ελπίζω να κατάλαβα καλά όμως, γιατί εσείς αναφερθήκατε για τις διαφορές των τιμών χονδρικής και λιανικής θέλετε εσείς να δημιουργήσετε σχετικές ανώτερες τριμές έτσι ώστε να λέμε ότι η λιανική τιμή να μην είναι τόσες φορές ε, η αντίστοιχη χονδρική. Και τέλος, μία από τις διαφάνειες που είδαμε έδειχνε και μου έκανε εντύπωση αυτό, αυτές τις τρευλώσεις των τιμών γύρω από το ανώτατο όριο. Αυτό δείχνει, θα έλεγα, κάτι. Είναι ένας δείκτης μιας κατάστασης η οποία προσωμιάζει σε καρτέλ. Διαρωτώ λοιπόν εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού να το εξετάσει αυτό. Γιατί μπορούμε να έχουμε αν θέλετε διορθωτικές συνταγές, διαρθρωτικές, μπορεί να χρησιμοποιούμε τα ανώτατα όρια τιμών, αλλά παρόλα αυτά ίσως και η αντίστοιχη Διεύθυνση Ανταγωνισμού να μπορεί να δει τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Μήπως πρέπει λοιπόν να το δούμε και αυτό. Σε όλες τις χώρες υπάρχει ένα συγκεκριμένος αριθμός ε, φυσικά ε, παροχέων και το να ε, διαμορφώνονται με κάπως ανορθόδοξο τρόπο οι τιμές, αυτό δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Το για. Πρόεδρε, όπως είπε και η συνάδελφος Έρτσογκ, Ξέρετε ότι ο κανονισμός τον οποίο περάσαμε στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο για το roaming, για την περιαγωγή, ήταν ε, βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δραστηριότητας απέναντι στον Ευρωπαίο πολίτη. Δεν ήταν κάτι το εύκολο λοιπόν, επί τη βάση της εμπειρίας που είχαμε και ε, εν μέρη επί τη της εν μέρη επιτυχούς συζήτησης που έγινε μέχρι σήμερα, μήπως μπορέσουμε να δράσουμε με περισσότερο θάρρος και με περισσότερη αποφασιστικότητα, έτσι ώστε να μπορέσουμε όλοι να καταστούμε εκ νέου πρωταγωνιστές της κατάστασης, ε, να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο ε, να είναι συμβατό με τις επιθυμίες των περισσότερων να περάσουμε σε μια ενιοποίηση των τιμολογήσεων σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι το νόημα της εσωτερικής αγοράς και εμείς είμαστε πολίτες οι οποίοι συνεχώς όλο και περισσότερο μετακινούμεθα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δυνατόν να πετύχουμε κάτι τέτοιο ή παραμένουν αυτά τα εμπόδια Ξέρουμε, ακούσαμε κα ήδη και κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περίοδου από πλευράς των κατανελητών ότι κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων μας έφεσαν στοιχεία τα οποία κανένας δεν μπόρεσε ε, να αντικρούσει σε σχέση με τις ανώτητες τιμές που δεν σέβονται σε καμία περίπτωση το πραγματικό κόστος και την απόσταση ανάμεσα στο κόστος το οποίο καλύπτει ο παροχέας και το κόστος το οποίο χρεώνει ο παροχέας. Λοιπόν, θα πρέπει κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων ανάμεσα στους καταναλωτές, τους παρεχείς και όλους τους εμπλεκομένους να δικαιολογηθεί αυτή η κατάσταση, να εξηγηθεί η κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έκανε αυτό, εξήγησε εν πάση περιπτώσει αυτό το θέμα του περιθωρίου κέρδους της αγοράς. Προφανώς και θα πρέπει να υπάρχουν κέρδη, προφανώς να υπάρξουν και νέοι παροχείς, αλλά όλα αυτά πρέπει να διευκρινιστούν. Θα ήθελα εγώ να μάθω ποια είναι η διαφορά του κόστους ανάμεσα στον παροχέα όταν παρέχει μια υπηρεσία στην Ιταλία, στη Γαλλία, στο Βέλγιο κτλ. Ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού του κόστους που τεκμηριώνει τη διαφορά του κόστους αυτού. Εγώ αντίθετα από τη συνάδελφο Χέρτσογκ είμαι τεμπέλα και έχω ένα τηλεφωνάκι μόνο, μόνο ένα και αυτό χρησιμοποιώ και πληρώνω εντελώς διαφορετικά τιμολόγια από χώρα σε χώρα. Λοιπόν, αυτή η διαφορά η οποία υπάρχει ανάμεσα στις μέγιστες χονδρικές τιμές και στη μέγιστη τελική τιμή λιανική στον χρήστη είναι τόσο μεγάλη και το είδαμε αυτό, πρέπει να καταλάβουμε γιατί έγινε αυτό. Ποιος ευνοείται από την κατάσταση αυτή, η αγορά. Για μου πείτε ότι ωφελούνται οι επιχειρήσεις ε, και δημιουργούνται λόγω αυτού του μεγάλου ποσοστού κέρδους νέες παροχές, ε, νέες υπηρεσίες κτλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζει η αγορά ε, και στην ουσία πράγματι δημιουργείται μια κατάσταση που μοιάζει με καρτέλ. Και τέλος, η τελευταία παρατήρηση την οποία θα ήθελα να κάνω. Οι προτάσεις οι οποίες γίνονται σχετικά με την υποστήριξη κάποιων <clears throat> τιμών συμβατών, να μπορεί κανείς με την ίδια ΣΥΜ να επιλέγει δύο παροχής. Αυτό τεχνικά είναι εφικτό. Το ρώτησε και η συνάδελφος Πινάδε Καστίγιο. Είναι λύσεις ενδιαφέρουσες ε, επιφανειακά, χρήσιμες για τον καταναλωτή. Αλλά μήπως έχουν τεχνικά κόστη τα οποία θα επιβαρύνουν ιδιαίτερα τη δραστηριότητα των παροχέων. Είναι δυνατόν να χαρακτηριστούν οι μέθοδοι αυτές ε, αναζήτησης ε, κάθε φορά του συμφεροτέρου παροχέα ουδέτερες σε επίπεδο τιμολογίων. Και τέλος, σημερίζομαι την θέση της Μπερέκ σχετικά με τις ανώτατες τιμές, τον καθορισμό των ανωτάτων ορίων και τη διατήρησή τους μέχρι τη στιγμή που θα είμαστε σίγουροι ότι η αγορά θα έχει πλέον ανοίξει και θα είναι ανταγωνιστική. Είναι μια εγγύηση αυτές οι ανώτατες τιμές. η κυρία Χόλ. Να ευχαριστήσω και, την, τον ΠΕΡΕΚ και την Κομισιόν για τις πολύ ενδιαφέρουσες αναλύσεις που ακούσαμε σήμερα το πρωί. Δύο ερωτήσεις έχω. Η Κομισιόν είπε ότι η νέα πρόταση θα βοηθήσει την πρόσβαση για τους παρόχους ε, υπηρεσιών, ε, για τους χειριστές των δικτύων. Ε, νομίζω όμως ότι πρόβλημα θα έχουν οι μικροί παροχοί υπηρεσιών, οι μικροί φορείς διότι συνήθω αυτοί δεν έχουν μεγάλες ε, μητρικές ε, εταιρείε ε, ή σημαντικές διασυνοριακές κοινοπραξίες όπως έχουν οι μεγάλοι φορείς. Όλοι γνωρίζουμε ότι στην πράξη δεν υπάρχουν συνθήκες ίσου ανταγωνισμού. μπορεί ε, να αποτύχει μια κλίση περιαγωγής ανάμεσα σε δύο χώρες ή ε, ένα SMS, ένα μήνυμα από κινητό να ε, απαιτήσει πολύ χρόνο για να παραδοθεί. Φαντάζομαι ότι πολλοί εδώ μέσα θα το έχουν ζήσει αυτό. Στην πρόταση αυτή λοιπόν δεν βλέπω τίποτα που να εξετάζει την ποιότητα των υπηρεσιών και που να επιδιώκει τη δημιουργία ίσων ε, συνθήκων ε, ανταγωνισμού όπου όλες οι κλήσεις ε, και όλα τα μηνύματα να έχουν την ίδια μεταχείριση. Και δεύτερον, όσον αφορά το θέμα του ανταγωνισμού, το βασικό πρόβλημα δεν είναι ότι ε, οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας δεν θέλουν ανταγωνισμό. Προτιμούν να έχουν μια ε, σιωπηρή συμφωνία, να μην έχουν ανταγωνισμό μεταξύ τους ε, και γι' αυτό οι τιμές να διαμορφώνονται κοντά στα ανώτατα όρια. Εγώ φοβάμαι ότι ακόμα και αν έχουν τη δυνατότητα παροχή τη δυνατότητας περιαγωγής οι επιχειρήσεις ε, δεν θα το επιλέξουν αυτό. Θα, ε, και το βλέπουμε αυτό και στην ε, αγορά ενέργειας με τους προμηθευτές αερίου και ηλεκτρικού που συνδυάζουν τις δύο προσφορές αυτές. Δεν βλέπω τίποτα στην προσφορά της Κομισιόν που να το εμποδίζει αυτό. Έτσι ουσιαστικά υπονομεύεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των ε, μεγάλων φορέων. Ευχαριστώ. Η κυρία Νίμπλερ, Αγγέλικα Νίμπλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τους ε, ομιλητές για την παρουσίαση του κανονισμού περί περιαγωγής. Ε, την εκτίμηση ότι ο κανονισμός του 2007 περί περιαγωγής ε, ήταν πολύ σημαντικός πολιτικά κανονισμός και είναι κάτι το οποίο ε, είχε σημαντική θέση και στις ε, ευρωεκλογές. Στηρίζω την πρόταση της κυρίας Χέρτσοκ. Ε, η επανεξέταση του θέματος αυτού να γίνει πριν το 2014 και όχι μετά τις ευρωεκλογές. Έχοντας κατά νου την ε, τον κανονισμό, τον υπάρχοντα κανονισμό και δίπλα μου κάθεται ο συνάδελφος Ρίμπιχ που τότε ήταν εισηγητής από πλευράς του Κοινοβουλίου. Ε, στο ε, Κοινοβούλιο είχαμε την ε, θέση γενικά ότι ήταν πολύ καλός ο κανονισμός αυτός και το θέμα ήταν αν ρυθμίσουμε τις τιμές περιαγωγής μήπως αυξηθούν οι εγχώριες τιμές. Αυτό είδαμε ότι δεν ε, συνέβη και ε, το δεύτερο ερώτημα ήταν ε, τα δεδομένα στην περιαγωγή. Τότε δεν είχαμε αρκετή κίνηση στον τομέα αυτόν ώστε να μπορούμε να συλλέξουμε επαρκή στοιχεία. Και γι' αυτό αναφέρθηκε στον κανονισμό ότι πρέπει να γίνει αναθεώρηση και ενδεχομένω να υποβληθούν νέε προτάσει αν υπάρξει σχετική ανάγκη. Όσον αφορά λοιπόν τη νέα πρόταση, Δεν έχω διαμορφώσει ακόμα θέση. Θα πρέπει να εξετάσω τα διαρθρωτικά μέτρα που ε, προβλέπει και η ΜΠΕΡΕΚ και η Κομισιόν. Γενικά όμως ε, βρίσκω καλή την προσέγγιση να ε, προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα της περιαγωγής όχι μόνο με ανώτετες τιμές αλλά και με διαρθρωτικές τροποποιήσεις. διότι θεωρώ πολιτικά κακή την ε, προσέγγιση με τις ανώτατες ε, τιμές, παρότι ήταν απαραίτητη τότε. Ε, πιο σωστό είναι να δώσουμε κίνητρα στην αγορά, να αυξήσουμε τον ανταγωνισμό. Βρίσκω λοιπόν γενικά καλή την προσέγγιση. Θα ήθελα και τον συνάδελφο από την ΠΕΡΕΚ και από την Κομισιόν θα ήθελα να ζητήσω από τους δύο συναδέλφους αυτούς ποια διαφορετικά μέτρα ε, θα πρέπει να ληφθούν, ε, ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στις δύο προτάσεις. Ε, και μία δεύτερη ερώτηση προς τον εκπρόσωπο του Μπέρεκ. Εάν έχουμε και εδώ αποδέσμευση θα έχουμε πιο εύκολη πρόσβαση στην αγορά νέων παρόχων υπηρεσιών. Ε, ο Μπέρεκ έχει λάβει παράπονα από φορείς που είπαν ότι δεν ε, μου δόθηκε πρόσβαση στην αγορά. Ε, το θέμα των καταναλωτών είναι άλλο, αλλά εμένα με ενδιαφέρει και, το, και η πλευρά των παρόχων. Και τέλος, βρίσκω καλή την πρόταση να έχουμε κατά νου όχι μόνο την εσωτερική αγορά, αλλά στον κανονισμό Ε, να συμπεριλάβουμε και ε, το, το κόστος που προκύπτει ε, εκτός Ευρώπης. Ο συνάδελφος Ρίμπιχ αναφέρθηκε στο θέμα αυτό εντός της Ευρώπης. Ε, αλλά ακούμε για λογαριασμούς πενταψήφιου σε ευρώ, μόνο και μόνο επειδή κατέβασε κάποιος μια εφημερίδα στο εξωτερικό. Ε, δεν θα πρέπει να κλείσουμε τα μάτια στο πρόβλημα αυτό. Γι' αυτό ε, ρωτώ την Κομισιόν, Ο Μπέρεκ ε, είναι υπέρ. Εσείς γιατί δεν έχετε ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Η συνάδελφος Τσίκαου. πολλοί από τους συναδέλφους οι οποίοι προελάλησαν θα συμφωνήσουν μαζί μου ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες εξετίμησαν δεόντως την, τον κανονισμό τον οποίο ψηφίσαμε για την περιαγωγή. Ήταν από τα λίγα τελικά μέτρα τα οποία λάβαμε σαν Ευρωπαίοι που έγιναν θετικά αντιληπτέ από τους πολίτες μας και οι οποίοι θεώρησαν ότι βελτιούται έτσι η καθημερινότητά τους. Ο κανονισμός λοιπόν, για, ο αρχικός κανονισμός για την περιαγωγή παρόλα αυτά δεν λειτουργήσε όπως θα έπρεπε και γι' αυτό προχωρήσαμε σε κάποιες τροποποιήσεις. Παρόλα αυτά τα τιμολόγια τα οποία εφαρμόζονται σήμερα νομίζω ότι είναι ιδιαίτερως υψηλά, είναι τα μέγιστα. Σε επίπεδο τιμής λοιπόν η κατάσταση πρέπει να αλλάξει. Διαπιστώσαμε ότι σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων ιδίω το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είδαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαμαρτυρίες από πλευράς των χρηστών λόγω των υψηλών λογαριασμών που κλήθηκαν να πληρώσουν. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο το κόστος του roaming και των μηνυμάτων να έρθει πιο κοντά στο πραγματικό κόστος της συγκεκριμένης υπηρεχίας. Οι τιμές των γραπτών μηνυμάτων και οι τιμολογήσεις των γραπτών μηνυμάτων θα πρέπει να ελεγχθούν πραγματικά στη σύνθεσή τους και ιδιαίτερα για τα γραπτά μηνύματα θα πρέπει να δοθεί μια προθεσμία για τον χρόνο άφηξης των μηνυμάτων αυτών γιατί πολλοί χρήστες ε, λαμβάνουν τα γραπτά μηνύματα όχι μετά από ώρες από τη στιγμή που απεστάλησαν αλλά μετά από ολόκληρες ημέρες. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρξει και ένα ευρωτιμολόγιο μετάβασης κατά τη διάρκεια του περάσματος στην περιαγωγή. Θα πρέπει να, οθωθεί, να προωθηθεί ένας ευρωπαϊκός κανονισμός ο οποίος φυσικά δεν θα πρέπει να είναι εχθρικός ούτε προς τον καταναλωτή ούτε προς τον παροχέα. Θα πρέπει να κατανοήσουμε σωστά τις διαφθρωτικές λύσεις τις οποίες προτείνει ο κανονισμός προς όφελος και του ανταγωνισμού και των καταναλωτών. Στο άρθρο 13 το οποίο δείχνει όπως βλέπετε τις συνθήκες για, την, για τον υπολογισμό των υψηλότερων αποδεκτών λιανικών τιμών. Βλέπουμε ότι οι όροι με τους οποίους έχουμε προχωρήσει στον υπολογισμό των τιμών και οι οποίοι θεωρούνται αποδεκτοί ε, μόνο από τη στιγμή κατά την οποία εφαρμοστούν πλήρως οι λεγόμενες διαρθρωτικές συνταγές οι οποίες δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως ακόμα. Μου φαίνεται λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξουν πιο συγκεκριμένες προτάσεις για τα επίπεδα των τιμών μετά από το 2015. Θα πρέπει να συλλέγονται τακτικά δεδομένα στοιχεία για τα τιμολόγια τα οποία εφαρμόζονται για όλους τους τύπους της περιαγωγής. Οι πληροφορίες αυτές δεν θα πρέπει να δίδονται μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και στο Κοινοβούλιο δίσκατέτος. Συνεπώς αυτό το οποίο ζητάμε εμείς είναι οι χρήστες να έχουν την δυνατότητα να επιλέγουν εναλλακτικούς παροχής και είναι απαραίτητο να υπάρξει μέγιστη δυνατή διαφάνεια και νομική βεβαιότητα για να το πετύχει τότε μόνο θα μπορέσουμε εμείς να δούμε αν μπορούμε ε, να αξιολογήσουμε σωστά τις περιαγωγές οι οποίες θα κοστίζουν και θα υπολογίζεται το κόστος τους με διαφορετικό τρόπο από ό,τι γίνεται σε επίπεδο εθνικό. Τότε μόνο θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε λοιπόν τη δυνατότητα αυτή ε, διαχωρισμένων, μάλλον διαφορετικών μορφών τιμολόγησης στο εξωτερικό από ό,τι σε εθνικό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια ζητήσαμε επανειλημμένα να υπάρξει μια προσαρμογή του κανονισμού αυτού και είπαμε ότι θα πρέπει να μειωθούν οι ανώτατες τιμές και είναι θετικό αυτό και επίσης είπαμε ότι είναι θετικό να δημιουργηθούν διαφορετικές συνθήκες που θα ευνοήσουν τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Όλες αυτές οι συνθήκες είναι απαραίτητες να υπάρχουν, είναι απαραίτητο να υπάρχουν στην επόμενη αναθεώρηση του κανονισμού. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Ε, ακούσαμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Ε, να ε, δώσω το λόγο ε, στην Κομισιόν για να προσπαθήσει να απαντήσει και κατόπιν θα ακούσουμε την Μπέρεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους ευρωβουλευτές για τα σχόλια. Δεν χρειάζεται καν να τα σχολιάσω για τα περισσότερα τα σχόλια. Θα προσπαθήσω να απαντήσω μόνο στις ερωτήσεις. Και ο διευθυντής του Μπερέκ θα απαντήσει πιο διεξοδικά στις ερωτήσεις που αφορούσαν την προσέγγιση του Φορέα Αριθμιστικών Αρχών. Εγώ θα επικεντρωθώ στα ζητήματα που αφορούν κυρίως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Δεκαστήγιο διαρωτήθηκε ποια είναι η ε, θεμελιώδης διαφορά μεταξύ των δύο προσεγγίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Μπερέκ. Και είπε ότι ίσως ε, ο Μπέρεκ δείχνει μια μεγαλύτερη δυσπιστία απέναντι στους φορείς εκμετάλλευσης, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πιο αισιόδοξη. Αυτό δείχνουν τα μέτρα που προτείνει. Ίσως να ισχύει αυτό ακούγοντας τον κύριο Φοντέιν και εμένα, ίσως αυτή την εντύπωση αποκομίσει κανείς. Πιστεύουμε ότι τα διαρθρωτικά μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχουν αντίκτυπο στην αγορά και ταυτόχρονα από τη στιγμή που το πιστεύουμε αυτό θα πρέπει να δώσουμε και εναύσματα στους φορείς εκμετάλλευσης για να εφαρμόσουν τις προτινόμενες λύσεις το συντομότερο δυνατόν. Χρειαζόμαστε επίσης ε, τους φορείς εγκατάλευσης, του παρόχους για να εφαρμόσουμε τα μέτρα. Δεν μπορούμε να έχουμε αφηρημένα κανόνες στις νομοθεσίες μας, γιατί σε τελική ανάλυση οι φορείς εκμετάλλευση είναι αυτοί που εμπράκτος θα εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη δική τους συμμετοχή. Γι' αυτό χρειαζόμαστε κίνητρα και ενάυσματα ώστε τα μέτρα αυτά να εφαρμοστούν όσο πιο γρήγορα και όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Και πιστεύουμε ότι ταυτόχρονα μαζί με τα μέτρα θα πρέπει να προτείνουμε και κάποια κίνητρα για την εφαρμογή τους. Και αυτή ήταν η ιδέα που δικαιολογούσε την άρση των ανώτατων τιμών. Και πριν το 2006, αν η αγορά μας δώσει ενδείξεις ότι η αγορά χάρη στα διαρθρωτικά μέτρα είναι ανταγωνιστική και φέρει αποτελέσματα ίσως ε, μετά το 2016 δεν χρειάζονται πια ανώτατα όρια τιμών. Βέβαια ταυτόχρονα, αν είμαστε υπεραισιόδοξοι και δεν δούμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, θα πρέπει ε, να δούμε στην αναθεώρηση αν κάποια διαρθρωτικά μέτρα χρειάζονται βελτίωση ή μήπως μερικά είναι τελείως αναποτελεσματικά. Αυτή την ισορροπία θα τη βρούμε. Αλλά για να εξασφαλίσουμε ωφέλη στους καταναλωτές θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και ενάψματα στη βιομηχανία για να καταστήσει την αγορά όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται. Ο κύριος Ρούμπιχ αναφέρθηκε στις τιμές περιαγωγής δεδομένων που θα μείνουν σε υψηλό επίπεδο για χρόνια ακόμη από ό,τι φαντάζομαι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ατυχής μεν, αλλά υπάρχουσα. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να επιληθεί αυτό το θέμα των υψηλών τιμών. Βέβαια, το θέμα είναι πώς θα ορίσουμε τα επίπεδα ανά τιμών περιαγωγής. Όπως είπα και προηγουμένως, θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία, ώστε και να αφήσουμε ελεύθερο τον ανταγωνισμό να αναπτυχθεί και ταυτόχρονα να έχουμε ένα μηχανισμό που θα τον ενισχύει, θα ενισχύει τον ανταγωνισμό, αλλά θα ορίζει ανώτατες τιμές που θα είναι σε τέτοιο επίπεδο ώστε να εξασφαλίζουν μια ελάχιστη προστασία και του καταναλωτή και του χρήστη. Βέβαια, αυτό θα λειτουργήσει εν μία νυχτή. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες διαφορές τιμών μεταξύ των ε, τοπικών δεδομένων και των δεδομένων της περιαγωγής και θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για να εξισωθούν αυτές οι διαφορές. Πάντως πιστεύουμε ότι με το συνδυασμό των μέτρων που προτείνουμε η εξομοίωση αυτή θα γίνει μάλλον γρήγορα. Κύριε Νίμπλερ, είπε ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε επιλογή για τους καταναλωτές και διαφάνεια. Με αυτό ακριβώ επιδιώκουμε και εμείς με την πρότασή μας. Τέθηκε και μία ερώτηση για τις μικρές χώρες και για το κατά πόσο η πρότασή μας δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση στις μικρές χώρες. Όσο ό,τι αφορά τις τιμές ελληνικής, όπως είπα και προηγουμένως με τους πίνακες που σας έδειξα, οι τιμές περισσότερο προσδιορίζονται από τις ρυθμιζόμενες ανώτατες τιμές. Δεν υπάρχουν δηλαδή μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών από αυτήν την άποψη. Ό,τι αφορά τις εναλλακτικέ προσφορές, εκεί υπάρχουν πιο μεγάλες διαφορές. Αλλά αυτές οι εναλλακτικές προσφορές στις διάφορες χώρες δεν προβλέπουν τιμές που είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις ε, προτινόμενες ανώτερες τιμές. Τώρα για τις μικρές χώρες και ιδιαίτερα για τους μικρούς ε, φορείς εκμετάλλευσης, για τους παρόχους. Και πώς θα φροντίσουμε με την πρότασή μας ε, να εξασφαλίσουμε συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού για τους μικρούς και για τους μεγάλους φορείς εκμετάλλευσης. Έχουμε καταρχήν τις ανώτατες τιμές χονδρικής. Αν θέλουμε να ενισχύσουμε τον ανταγωνισμό, χρειαζόμαστε τιμές χονδρικής για όλους τους φορείς εκμετάλλευσης, και τους μικρούς και τους μεγάλους, αλλά και τους ε, δυνάμει νέους φορείς, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν ε, ενδιαφέρουσες προσφορές Λενικής και ενδιαφέρουσες τιμές Λενικής. Αυτή την άποψη, οι ανώτατες τιμές ε, ε, χονδρικής που προτείνουμε είναι αρκετά αυστηρές και δεν προσανατολίζονται τόσο στο κόστος. Και με αυτές τις ανώτατες τιμές χονδρικής και οι μικροί φορείς εκμετάλλευση αλλά και οι νέοι, οι νέοι εισερχόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν τους ε, καθιερωμένου ή μεγαλύτερου φορεί εκμετάλλευσης. Ο κύριος Μπέλετ ρώτησε για την κατάσταση στις άλλες χώρες, Ηνωμένε Πολιτείε και άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας απαντήσω, για τον το λόγο ότι η αγορά περιαγωγής ρυθμίζεται μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς συγκεντρώνουμε στατιστικά στοιχεία από τους φορείς εκμετάλλευσης, αλλά σε άλλες χώρες του κόσμου δεν υπάρχει τόσο συστηματική συγκέντρωση στοιχείων. Υπάρχουν κάποιες εμπορικές συμφωνίες, αλλά δεν ξέρω αν ο συνάδελφο από τον Μπερέκ έχει πληροφορίες για τις τιμές σε άλλε χώρε του κόσμου, αλλά εγώ τέτοιε πληροφορίες δεν διαθέτω. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος για τις πωλήσει προϊόντων γυναικείων τσαντών. <laughs> Ελπίζω να μην βλάψουμε την αγορά γυναικείων τσαντών με την πρόταση αυτή, αλλά ακόμη και γίνει αυτό φαντάζομαι ότι θα αναπτυχθούν άλλα προϊόντα που θα ανταποκρίνονται στη ζήτηση. Αν αυτό συμβεί με τον κανονισμό της περιαγωγής, αναπτυχθούν τέτοιες αγορές, θα χαρούμε ιδιαίτερως. Ο κύριος Λάμπερτ ρώτησε αν είχαμε διαβουλεύσεις με οργανώσεις καταναλωτών πριν καταθέσουμε την πρότασή μας ή πριν ε, προβούμε στις δημόσιες διαβουλεύσεις. Είχαμε συζήτηση με όλους τους ε, ε, φορείς και ενδιαφερόμενους και τη βιομηχανία και τις οργανώσεις καταναλωτών. Ήταν ευρύτατες οι διαβουλεύσεις και κάτι που δείχνει την περιπλοκότητα το, της αγοράς είναι ότι όλοι και οι ενδιαφερόμενοι και η βιομηχανία και οι καταναλωτές ενδιαφέρονται για την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ανταγωνισμού στην αγορά περιαγωγής. Το παράδοξο όμως είναι ότι δεν ε, υπέβαλαν συγκεκριμένες προτάσεις. Ούτε και εμείς ε, είχαμε τότε συγκεκριμένες προτάσεις για τα διαρθρωτικά μέτρα. Ούτε η βιομηχανία υπέβαλε κάποια συγκεκριμένη πρόταση. Και από ό,τι ακούσαμε από τον Μπερέκ, ίσως η βιομηχανία δεν πιστεύει ότι υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση εκτός από μια επιλεκτική εφαρμογή. Ήταν κάπως αφηρημένες οι συζητήσεις αρχικά και μόνο μετά την ολοκλήρωση των δημόσιων διαβουλεύσεων καταρτήσαμε τη δική μας πρόταση, έχοντας ε, εξετάσει όλα τα επιχειρήματα και θεωρώντας ότι είναι και η πιο δόκιμη λύση. Οι καταναλωτές, οι οργανώσεις καταναλωτών, πριν την υποβολή της πρότασης δεν είχαν ε, εκφέρει σχόλια. Τώρα έχουν λάβει γνώση και περιμένουμε τις αντιδράσεις τους. Φυσικά οι καταναλωτές ενδιαφέρονται για συμφέρουσες συμφωνίες και πακέτα που θα εξασφαλίσουν καλή ποιότητα υπηρεσιών και χαμηλές τιμές. Οπότε η έμφαση που δίνουν σε απαντήσεις τους οι οργανώσεις καταναλωτών στις δημόσιες διαβουλεύσεις είναι, δίνεται στην ανάγκη ε, συνέχισης της ρύθμισης των τιμών. σε ό,τι αφορά τον πιθανό σχηματισμό καρτέλ στην αγορά και αν έχει ξεκινήσει κάποια έρευνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο μετά το 2000. Τότε είχαμε κάνει μια σχετική έρευνα για την περιαγωγή και απέβη άκαρπη. Και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο καρτέλ αν το ήξερα θα το κατήγγειλα στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού για να το ελέγξει. Πάντως, ίσως, ο κανονισμός με τις ανώτερες τιμές ίσως δημιουργήσει τη δυνατότητα στους, καταναλ... στους φορείς εκμετάλλευσης να συνεργαστούν, ίσως όχι καταλήγοντα στις συμφωνίε, αλλά ίσω ε, υιοθετώντα μια προσέγγιση. Βλέπουν ποιο είναι, ποια είναι η ενότατη τιμή και γνωρίζουν ποιε είναι οι τιμέ. οπότε αυτή την άποψη είναι εύκολο να καταλήξουν οι φορείς ε, εκμετάλλευση στο συμπέρασμα ότι αν υποβάλλω μια τιμή ε, στο επίπεδο τη ανώτατη τιμή, ή λίγο χαμηλότερη, τηρούμε τον κανονισμό και μπορούμε να εξασφαλίσουμε και το κέρδος μας το γεγονός ότι οι τιμές περιστρέφονται γύρω από την ανώτατη τιμή οφείλεται και στον κανονισμό. Και γι' αυτό το λόγο ίσως θα πρέπει να αναζητήσουμε και εναλλακτικέ λύσεις. Ρωτήθηκε και το ποιο είναι το περιεχόμενο των διαρθρωτικών μέτρων και ποιες είναι οι διαφορές μας με τον Μπερέκ. Θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω για μια ακόμη φορά τι είναι αυτά τα διαφορετικά μέτρα. Υπάρχουν δύο προτάσεις. Υπάρχει καταρχάς η υποχρέωση εισδοχή στην χοντρική αγορά, εναλλακτική ε, παροχής, οποιοδήποτε θέλει να παρέχει υπηρεσίες περιαγωγής θα έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες περιαγωγής των βασικών χρηστών. Αυτό είναι κάτι των βασικών παροχείων, συγγνώμη. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς προτείνουμε και πρέπει να γίνει δεκτό. Και το άλλο θέμα είναι τη λεγόμενη απελευθέρωση των υπηρεσιών ή ε, αποδεσμοποίηση των υπηρεσιών στον τομέα της περιαγωγής. Προσπαθήσαμε να δούμε σε τι αυτό ωφελεί στους χρήστες από τη μία και στους παροχείς από την άλλη για τους καταναλωτές και ξεκινώ από αυτούς, τους δίνει τη δυνατότητα, το unbundling, η αποδεσμοποίηση, να προσπαθήσουν να εξετάσουν τις διάφορες προτάσεις οι οποίες προσφορές που υπάρχουν, διατηρώντας όμως τον δικό τους παροχέα για το, ε, για το εσωτερικό της αγοράς στην οποία κινούνται. Και για τους παροχείς πιστεύουμε ότι η αποδεσμοποίηση είναι απαραίτητη γιατί και σε σχέση με το πρώτο μέτρο δίνει τη δυνατότητα στους παροχείς να προτείνουν με μονομένες υπηρεσίες περιαγωγής. Πολλές φορές οι παροχείς οι οποίοι θέλουν να δίνουν υπηρεσίες μόνο σε επίπεδο περιαγωγής δυσκολεύονται να μπουν στις αγορές. Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα της απελευθέρωσης, της αποδεσμοποίησης, δύσκολα ξεφεύγει κανείς από τον παροχέα της, ε, που χρησιμοποιεί σε εσωτερικό, σε εθνικό επίπεδο. Γι' αυτό ακριβώς τα μέτρα αυτά αποδεσμοποίησης θεωρούμε ότι είναι απαραίτητα. Υπήρξαν και κάποιες άλλες ερωτήσεις σχετικά με την ποιότητα των παρεχωμένων υπηρεσιών και τις καθυστερήσεις στην παράδοση των γραπτών μηνυμάτων. Νομίζω ότι αυτά καλύπτονται από τον ενισχύ κανονισμό. Γενικότερα η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας και στον τομέα της περιαγωγής και στον τομέα της εθνικής υπηρεσίας είναι κάτι το οποίο καλύπτεται από τον κανονισμό πλαίσιο και θα πρέπει οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές των τηλεπικοινωνιών να παρακολουθούν κατά πόσον υπακούν και είναι συμβατές οι συμπεριφορές των εταιριών παροχέων με τον κανονισμό. Αίσθησή μου είναι ότι μπορώ να κλείσω, ζητώ συγγνώμη αν κάτι ε, μου διέφυγε, είμαι στη διάθεσή σας πάντως. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Αν υπάρξουν περισσότερες τεχνικές ερωτήσεις, ίσως ε, ο εκπρόσωπος της Μπερέκ θα μπορέσει να συμπληρώσει αυτά τα οποία είπατε. Εγώ δεν θα επαναλάβω τα διαφορετικά θέματα τα οποία ακούστηκαν μέχρι τώρα. Θα ήθελα να έλθω στη συμφωνία που υπάρχει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Μπερέκ γύρω από όλα αυτά τα θέματα. Υπάρχουν ίσως κάποια θέματα στα οποία έχουμε κάποιες διαφορές, αρκετά ίσως, αλλά παρόλα αυτά στα βασικά νομίζω υπάρχει μια συμφωνία. Ξέρετε ότι όταν υπάρχουν δύο οικονομολόγοι να συζητούν σε μία αίθουσα εκφράζονται τρεις απόψεις συνήθως. Το ίδιο ισχύει και με τους περιαγωγικούς δεν υπάρχει μία ενιαία λύση η οποία να είναι απόλυτα καλύτερη από όλες τις υπόλοιπε προσφερόμενες. ω εκ τούτου είναι λογικό να υπάρχουν διαφορετικέ απόψεις. Υπάρχουν τέσσερα θέματα τα οποία θα ήθελα, στα οποία θα ήθελα να σταθώ και στα οποία διαφέρομαι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρώτο, ο βαθμός εμπιστοσύνης τον οποίο έχουμε αναπτύξει στην αποτελεσματικότητα ε, της μεθόδου της ε, απελευθέρωσης αποδέσμευσης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι μια σημαντική στρατηγική. Εμείς έχουμε επιφυλάξεις γύρω από αυτό. Είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει σωστά μια τέτοια μέθοδος. Δεν ξέρουμε επίσης και ποια θα είναι η συμπεριφορά των καταναλωτών. Δεν είναι ότι είμαστε κατά της ύπαρξης περισσότερου ανταγωνισμού ή περισσότερης επιλογής ε, του καταναλωτή. Αλλά είμαστε επιφυλακτικοί ε, για τα συγκεκριμένα ωφέλη. Το δεύτερο θέμα, όπου διαφέρουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι οι ανώτατες τιμές λιανικής. Πιστεύουμε ότι τα όρια αυτά θα πρέπει να τίθενται, έτσι όπως είναι τα πράγματα, έτσι ώστε να υπάρχει έλογο κέρδος από πλευρά των παροχέων. Συμφωνούμε επίσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι θέλει να διευκολύνει την είσοδο των νέων αν θέλετε παροχέων. Και γι' αυτό θα πρέπει να είναι κανείς λίγο πιο γενικό, γενναιόδωρος σε σχέση με τις ανώτατες τιμές. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο ανταγωνισμός θα καταργήσει την ανάγκη η οποία υπάρχει για τον καθορισμό των ανωτάτων τιμών. Εδώ λοιπόν είμαστε επιφυλακτικοί. Πιστεύουμε ότι τα περιθώρια είναι σε επίπεδο το οποίο θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες των επιχειρήσεων και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφόσον πράγματι σταθεί γενναιόδορη σε σχέση με τον καθορισμό αυτών των ανωτάτων τιμών τότε θα μπορέσουμε να υποστατεύσουμε τα συμφέροντα των καταναλωτών σωστότερα. Συνδεόμενο με το θέμα αυτό είναι και το θέμα της κατάργησης των ανωτάτων τιμών και της διάρκειας ισχύω των υπαρχουσών ρυθμίσεων και κατά πόσον οι δυνάμεις της αγοράς δείχνουν ότι είναι ικανές να απομακρύνουν, να καταργήσουν την ανάγκη ύπαρξης αυτών των, των ποσοστών κέρδους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να κάνει κάποιες ε, ε, αλλαγές εφόσον βέβαια ε, δεν υπάρχει πλέον ανάγκη διατήρησης των ανωτάτων τιμών. Εμείς προσπαθούμε να πούμε ότι θέλουμε να διατηρηθούν οι ανώτατες τιμές εφόσον δεν έχουν υπάρξει αποδείξεις για την αλλαγή της κατάστασης στην αγορά. Στα τελευταία στοιχεία τα οποία θα δημοσιεύσουμε σε, σε επόμενες εβδομάδες βλέπουμε δυστυχώς ότι υπάρχουν κάποιες ε, αυξήσεις ε, στον τομέα ε, των λεγόμενων μη ρυθμιζομένων εναλλακτικών τιμολογήσεων. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν καλύτερες τιμές για τους καταναλωτές, αλλά οι στατιστικές μέχρι τώρα δεν το δείχνουν οι τιμές των εναλλακτικών παροχέων είναι ανώτερες συνήθως από τις τιμές τις οποίες προσφέρουν οι, οι βασικοί παροχείς. Και τέλος θα ήθελα να υπογραμμίσω για μια ακόμη φορά το θέμα το οποίο ανέφερε ο κ. Φοντέιν στο τέλος της ομιλίας του, της πρότασης την οποία κάνουμε για τη διεύρυνση της δυνατότητας προστασίας του καταναλωτή και εκτός Ευρώπης θα θέλαμε να υπάρξει μείωση του κόστους της περιαγωγής και εντός και εκτός Ευρώπης. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια της νομοθετικής ρύθμισης της εσωτερικής αγοράς. Εμείς πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να ελέγξουμε τα ποσοστά των επιχειρήσεων έτσι ώστε ε, να είναι σε θέση οι επιχειρήσεις ε, να προειδοποιούν τους καταναλωτές όταν εκτίθενται σε υπερβολικές χρεώσεις εντός και εκτός Ευρώπης. Αυτό θα ήταν κάτι το καλό να μπορούσαμε να το προτείνουμε. Αυτή είναι η τομή στους οποίους λοιπόν ίσως θα ελαφρώσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάρα πολύ σύντομα να έλθω σε κάποιες από τις συγκεκριμένες ερωτήσεις που τέθηκαν από τα μέλη σας σχετικά με τον ανταγωνισμό και επανέρχομαι σε αυτά τα οποία έλεγα πριν λίγο, εμείς μπορούμε να νομοθετήσουμε σαν παράδειγμα ότι οι τιμές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν ένα επίπεδο. Αυτό είναι όμως κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους παροχείς. Εμείς καθορίζουμε σωστά τις τιμές αλλά δεν βελτιώνεται ο ανταγωνισμός, οι συνθήκες ανταγωνισμού. Λοιπόν, αν δεν έχουν εμπορικό συμφέρον οι παροχείς να ανταγωνιστούν θα το κάνουν. Αν δεν έχουν δεν θα το κάνουν πάρα πολύ απλά. Αυτό συνδέεται λίγο και με τις ανησυχίες μας σχετικά με τα μέτρα για την απελευθέρωση, την αποδεσμοποίηση. Προφανώς όταν μας ζητείτε να προσφέρουμε την αποδεσμοποίηση θα το κάνουμε, δεν υπάρχει αμφιβολία. Το θέμα είναι τι επιπτώσεις θα υπάρχουν στους καταναλωτές, θα χρησιμοποιήσουν τις νέες αυτές δυνατότητες έτσι ώστε να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές οι οποίες να είναι πιο ελκυστικές. Αν όχι τότε τα μέτρα δεν θα έχουν ιδιαίτερα μεγάλη θα έλεγα σημασία. Για τις τιμές ε, των ε, δεδομένων ε, στην Αυστρία κυρία Ρούμπικ το πρόβλημα δεν είναι βέβαια μόνο το να κατεβάζετε ταινίες στο κινητό σας το θέμα είναι ότι δεν μπορείτε να βάλετε μπρο το smartphone σας απλά μερικές φορές σε ορισμένες χώρες, γιατί αυτό μπορεί να σας κοστίσει πολύ. Γιατί πάρα πολύ συχνά κατεβάζουν οι χρήστες δεδομένα χωρίς να το καταλαβαίνουν, χωρίς να παίρνουν είδηση τι γίνεται μέσω των smartphones Πρέπει λοιπόν οι τιμές αυτές να μειωθούν ακόμα περισσότερο σε επίπεδα τα οποία να είναι πολύ πιο κοντά στα εθνικά επίπεδα έτσι ώστε να μπορούν οι χρήστες να χρησιμοποιήσουν τα smartphone που έχουν με αποτελεσματικότερο τρόπο. Τιμές και κόστος. Εμείς ε, δημοσιεύσαμε κάποια στοιχεία στην έκθεσή μας τον μήνα Δεκέμβριο για το κόστος ε, και τις τιμές των περια... της, η αξιολόγηση των στοιχείων που έχουμε στη διάθεσή μας και τα μοντέλα κοστολόγησης που έχουμε ίσως να είναι λίγο ξεπερασμένα. Αλλά το κόστος, το υποβόσκον αν θέλετε για την παροχή των, ε, των υπηρεσιών περιαγωγής δεν διαφέρει και πάρα πολύ από τις άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες και υπάρχουν δυνατότητες για τη μείωση του κόστους όπως ακριβώς το έχουν κάνει και σε εθνικό επίπεδο οι, α, οι παροχείς οι οποίοι κερδίζουν αρκετά. Για τις μικρότερες χώρες πράγματι για τις υπηρεσίες περιαγωγής όπως επίσης και για άλλες υπηρεσίες οι καταναλωτές στις μικρές χώρες, όχι σε όλες αλλά σε πολλές, δεν τα καταφέρνουν τόσο καλά από πλευράς τιμολόγησης από σε μεγάλες χώρες. Για τους μικρούς παροχής ακούσαμε ότι προστατεύονται από τις νέες προτινόμενες ε, ε, ανώτατες τιμές. Οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν χρειάζονται την προστασία αυτή, μπορούν από μόνες τους να προστατευτούν και να κάνουν συμφωνίες που τις συμφέρουν. Οι μικροί παροχείς δεν το έχουν αυτό και ωφελούνται. Αντίθετα με τον καθορισμό των τιμών της Λιανικής θα ήθελα να πω ότι σε αυτή τη φάση δεν προβλέπω να καταστεί γρήγορα άχρηστη δυνατότητα καθορισμού τιμών στην χονδρική αγορά. Νομίζω ότι εξακολουθεί η ρύθμιση των τιμών στον τομέα αυτό να είναι απαραίτητη για αρκετό καιρό. Σχετικά με τις τσάντες των γυναιτών δεν καταλαβαίνω και πάρα πολλά πράγματα, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να προσβλέπουμε σε μία φάση, όχι πολύ μακριά στο μέλλον, όπου θα είναι προς το συμφέρον το εμπορικό των επιχειρήσεων να προσφέρουν τιμολόγια ευρωπαϊκά, να πληρώνει κανείς τα ίδια όπου και αν είναι στην Ευρώπη και αυτό θα διευκολύνει φυσικά την ανάγκη που υπάρχει σήμερα να κουβαλάει κανείς μεγάλες τσάντες για τον κύριο Λάμπερτ και για τη σχέση ανάμεσα στις φονδρικές και, νομικές τιμές, και ελιανικές συγγνώμη, τιμές. Πάνω κάτω εδώ έχω απαντήσει. Νομίζω ότι σε μια διαγωνιστική αγορά μπορεί κανείς να περιμένει την λιανική αγορά να είναι κοντά θα έλεγα να είναι βασισμένη στις ρυθμίσεις ε, με τις οποίες λειτουργεί η χονδρική αγορά. Και εκεί υπάρχει δυνατότητα μείωσης ε, του περιθωρίου ανάμεσα στη λιανική και τη χονδρική για την επιλογή των διαφορετικών μέτρων τώρα, όπως είπε ο κ. Φοντέιν στην παρατήρησή του. Έχουμε κάνει αρκετή δουλειά στον τομέα αυτό τον τελευταίο χρόνο. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν κάποια διαφορετικά μέτρα ικανοποιητικά, αλλά όχι να αντικαταστήσουμε όμως ε, να αντικαταστήσουμε τις ανώτατες τιμές. Νομίζω ότι μπορούμε να εξαρτηθούμε εν μέρη από τις διαφορετικές τιμές, από, τις, από τα διαφορετικά μέτρα και εν μέρη από τον καθορισμό των ανωτέρων τιμών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα είναι εύκολο να εφαρμοστεί και δεν θα κοστίσει ιδιαίτερα. Θα πρέπει να υποστηριχθεί βέβαια από, μεγάλη, από το μεγάλο ποσοστό της αγοράς, γιατί χωρίς την υποστήριξη της αγοράς τα διαφορετικά μέτρα από μόνο τους δεν θα ε, βοηθήσουν πολύ. Κυρία Νίμπλα, ε, μας μίλησε για την πρόσβαση στο δίκτυο. Υπάρχουν εταιρείε οι οποίες ζητούν συνεχώς να μπουν στα δίκτυα ε, κάλοτε το πετυχαίνουν, άλλοτε όχι. Οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται από τις ρυθμιστικές αρχές, αλλά λαμβάνονται με βάση την εμπορική λογική θα έλεγα. Δεν είναι κάτι το οποίο οι ρυθμιστικές αρχές ασχολούνται ιδιαίτερα, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο ρυθμίζεται πάρα πολύ απλά και θα... δεν μπορούμε σαν ρυθμιστικές αρχές να κάνουμε πολλά πράγματα γύρω από αυτό, οπότε δεν έχει και νόημα να τα συζητάμε ιδιαίτερα. Αυτά, αν ξέχασα κάτι, στη διάθεσή σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά και τους τρεις προσκεκλημένους μας. Ένας έπρεπε να μας εγκαταλείψει νωρίτερα. Να ευχαριστήσω και εσάς για τις πολλές ερωτήσεις, τις παρεμβάσεις σας. Νομίζω ότι ήταν χρήσιμο ε, που συζητήσαμε το θέμα αυτό έτσι συγκεντρωμένα. Νομίζω ότι θα ε, διευκολύνει αυτό τις εργασίες μας. Σήμερα το απόγευμα θα πρέπει να αλλάξουμε τη σειρά ε, ανάμεσα σε δύο θέματα. Το 4 και το 6 θα αντιστραφούν διότι θα θα καταφτάσει αργότερο ο προσκεκλημένος μας για το σημείο 4. Ε, γι' αυτό λοιπόν θα εξετάσουμε πρώτα το σημείο 6 και το 4 θα μπει στη θέση το 6. Ωραία, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι, τα λέμε αργότερα.